Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Point of order. Adam. διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω στους συναδέλφου αυτό που είπε η γαλλική κυβέρνηση για την ψηφοφορία που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περασμένη Πέμπτη ε, σε σχέση με τους Ρωμά. Το γαλλικό κοινο... Η γαλλική κυβέρνηση καταπατά τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα μπορούσαμε να πούμε. Μας, ε, μας ε, κατηγορεί για πολιτικαντισμούς και μας λέει ότι δεν έχουμε τέτοια δικαιώματα και ότι παραβιάζουμε ή μάλλον περιφρονούμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες ε, για λόγους πολιτική, της δικής μας πολιτικής. Χαίρομαι που βρίσκεται εδώ η κυρία κανονες για λογους τη Το Σαββατοκύριακο η γαλλική, ο γαλλικός τύπος απεκάλυψε μια εγκύκλιο που ε, παραβιάζει όλα όσα είπατε εσείς κυρία Επίτροπε και οι συναδελφοί σας στη γαλλική κυβέρνηση γιατί μιλάει ρητά για την ε, αποβολή, για την εκδίωξη των ε, καταβλισμών των Ρωμά και μιλάει μόνο για αυτούς. Έτσι, η γαλλική κυβέρνηση, η οποία από την περσμένη πέμπτη μας εξηγεί ότι πρέπει οι Ρουμάνοι να μάθουν να γίνουν ε, Ευρωπαίοι πολίτες, θα ήθελα να στραφώ στους, Ρωμα... στους Ρουμάνους και Ούγγρους συναδέλφους πρέπει να μάθει η γαλλική κυβέρνηση σε αυτούς τους ανθρώπους να είναι ε, Ευρωπαίοι πολίτες. Υπάρχουν όρια θα έλεγα για οποιαδήποτε κυβέρνηση και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει και κάποια κοινοβουλευτική αλληλεγγύη. Γνωρίζω κύριε Πρόεδρε και ότι και οι συντονιστές θα ασχοληθούν με το θέμα, όμως θα ήθελα κάτι επιγόντως να ακούσουμε τις κυρίες Ρέντιν και Μάλστρομ για να μάθουμε ακριβώς τι ακριβώς τους είπε η γαλλική κυβέρνηση και για να μάθουμε όλοι τα όσα λέει αυτή η εγκύκλωση την οποία θα δώσω και σε εσά κύριε Πρόεδρε και στην κυρία Μάλστρομ. Το σημειώνουμε, σημειώνουμε τα σχόλιά σας κύριε Βερζάτ. Έγινε η ψηφοφορία στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα και θα δούμε ποιο θα είναι το follow-up, η συνέχεια που θα δώσουμε κατά τους συντονιστές. Προτείνω λοιπόν κυρία Ζερζά να προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη και να ακούσουμε την κυρία Σεσίλια Μάλστρομ, την Επίτροπο. Μετά την κυρία Μάρστρομ λοιπόν θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη, θα την ολοκληρώσουμε και μετά στους συντονιστές θα δούμε τι θα γίνει με τη συνέχεια της ψηφοφορίας. Τη συνέχεια θα δώσουμε στην ψηφοφορία. για την απέλεση των Ρώμα και τις απαντήσεις που μας έδωσε η γαλλική κυβέρνηση. Όπως είπαμε, όπως συνήθως, θα συνεχίσουμε πρώτον με την έγκριση της μερίσιας διάταξης. Αντιρρήσεις εγκρίνεται. Δεύτερον, όσον αφορά τις ανακοινώσεις. Ένα θέμα για μια προθεσμία ε, υποβολή τροπολογιών. Μετά από πρόταση του εισηγητή, εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι η προθεσμία ε, υποβολής τροπολογιών που αφορά το πακέτο χωρίς ασύλου ε, ε, που εισηγητή είναι ο συνάδελφος κύριος Μωράες ανοίγει σήμερα και θα κλείσει η προθεσμία αυτή το μεσημέρι της 29 Σεπτεμβρίου. Μία μέρα μετά την υποβολή της, του σχεδίου έκθεσης, 29 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι λοιπόν. Η έκθεση ήδη υπάρχει σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, μπορεί να έρθετε σε επαφή με την γραμματεία της ε, ομάδας. Λίμπε. Της Επιτροπής, συγγνώμη. Και τώρα περνάμε στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων, των προηγούμενων συνεδριάσεων της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Υπάρχουν εδώ. Αν δεν υπάρχει κάποια παρατήρηση για τα πρακτικά, θεωρούμε ότι έχουν εγκριθεί. Οπότε, περνάμε στο τέταρτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις και τις μελλοντικέ προτεραιότητες στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Οπότε, επ' αυτού, έχουμε την χαρά για μία ακόμα φορά να έχουμε μαζί μας την Επίτροπο κυρία Σεσίλια Μάλστρομ, η οποία θα μας κάνει μία επισκόπηση των πρόσφατων εργασιών και των προτεραιοτήτων στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μία εξαιρετική πρακτική, ε, την οποία εφαρμόζουμε ήδη από τις αρχές Μαΐου και έχει αποδειχθεί όχι μόνο σημαντική αλλά και χρήσιμη γιατί ε, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δείχνουμε τη δουλειά μας. Καλώς ορίσατε κυρία Επίτροπε. Θα σας ακούσουμε και μετά θα περάσουμε στη συζήτηση. Η κυρία Μάλστρομ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω. Ε, Είχαμε ξανασυναντηθεί, όπως είπε και ο Πρόεδρος, το Μάιο και έκτοτε έχουν συμβεί πολλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας πω τι έχει συμβεί και επίσης τι ε, υπάρχει στο πρόγραμμα των εργασιών μας του φθινοπόρου. Χαίρομαι πολύ που η συνεργασία μας έχει εξελιχθεί με τόσο επικοδομητικό και θετικό τρόπο ε, και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με αυτόν τον τρόπο και στο υπόλοιπο της θητείας. Ε, φυσικά και δεν θα μπορέσω να αναφερθώ σε όλα τα θέματα. Έχουμε όμως αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας και θα μπορέσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ξεκινώντας με αυτά τα οποία έγιναν τους τον τελευταίο μήνα, θα ξεκινήσω από την πολιτική της μετανάστευσης. Πριν ε, ακριβώς τις διακοπές, ε, η Επιτροπή υιοθέτησε δύο νομοθετικές προτάσεις για θέματα νόμιμης μετανάστευσης. Είναι για την ε, ενδοετερικές μεταθέσεις και τις εποχιακούς εργάτες. Η πρώτη αφορά μια νέα ταχεία διαδικασία για ειδικούς εργαζόμενους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, μετατίθενται προσωρινά στα γραφεία μιας εταιρείας ενός κράτους μέλους. Όσον αφορά τους εποχιακούς εργαζόμενους θα υπάρξουν ειδικέ διατάξεις για ε, μια δυνατότητα μετάβασης μέχρι 6 μήνες και πολλαπλές εισόδους. Και βεβαίως υπάρχουν και ειδικοί, ε, ειδικές για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών πρακτικών. Στόχος ε, της έγκρισης αυτός είναι να προωθηθεί η κοινή μεταναστευτική πολιτική και να συμπληρωθούν και άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Επί του ασύλου, μετά τον έγκριση, τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Γραφείου Στήριξης Ασύλου το Μάιο. Ε, θέλουμε το 2011 να υπάρχει αυτό το γραφείο συμπεριλαμβανομένου και του εκτελεστικού διευθυντή του φέτος ελπίζουμε. Μια άλλη ε, σοβαρή εξέλιξη που είδαμε τους τελευταίους μήνες είναι η ενασχόληση της Επιτροπής ε, σε πολύ πικοδομητικό διάλογο με τις ελληνικές αρχές που ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε χειροπιαστές βελτιώσεις της ελληνικής πολιτικής στον τομέα της παροχής ασύλου. Έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης ε, στα χέρια μας που υπέβαλε ε, η ελληνική κυβέρνηση και σε λίγο καιρό θα επισκεφθώ την Ελλάδα για να συζητήσω την εφαρμογή του και τις λεπτομέρειές του. Για το ΣΥΣ2 και παρά κάποιες δυσκολίες, Περάσαμε το Μάρτιο το πρώτο, την πρώτη σημαντική δοκιμασία και αυτό δείχνει ότι η ανάπτυξη μπορεί να αποτελέσει βάση και αυτό με, βάση κάποια κοινή αξιολόγηση από το Συμβούλιο, οι υπηρεσίε Επιτροπή έχουν ξεκινήσει λεπτομερεί διαπραγματεύσει με τον ανάδοχο και θα επιβάλλουν συγκεκριμένε προτάσει στο ε, Συμβούλιο Τζάι του Οκτωβρίου. Και φυσικά και εσεί θα τηρήσετε τακτικά ενήμεροι για τη διαδικασία αυτή τι ερχόμενε εβδομάδε. Όσον αφορά τη ΦΙΖΑ, πολλά έχουν γίνει Ο κώδικα θεωρήσεων που ισχύει από την 5η Απριλίου φέτος εξυγχρονίζει όλη τη σχετική νομοθεσία για την επεξεργασία και την πρόθεση των αιτήσεων για θεωρήσεις ε, και έχει εξυγχρονιστεί μέχρι το τέλος Μαΐου. Η Κομισιόν είχε εγκρίνει μια ε, νομοθετική πρόταση η απελευθέρωση θεωρήσεων στην Αλβανία και στους πολίτες Αλβανίας και Βοσνίας Ρεκοβίνης και έκτοτε ε, έχω μια αξιολόγηση και νομίζω ότι την έκθεση την έχετε ήδη λάβει. Η πρόταση για τη μεταφορά της Ταϊβάν στο θετικό κατάλογο επίσης εγκρίθηκε από την Κομισιόν στις 15 Ιουλίου. Η Ταϊβάν έχει επίση δώσει ε, ε, εκφράσει θελησή να χορηγήσει ελεύθερη θεώρηση σε όλου του ευρωπαίου πολίτε. Θα έχουμε... Έχουμε επίση ρυθμίσει με τη Βραζιλία. Θα υπογραφεί με το τέλο του χρόνου συμφωνία και θα υπάρχει πλήρη ελευθερία και από τι δύο πλευρέ. Μια συμφωνία διευκόλυνση θεωρήσεων με τη Γεωργία. Τον Οκτώβριο υπάρχει μια αρχική συμφωνία, αλλά ε, υπάρχει και υπάρχουν και άλλε διαταγές για το TFTP. Για μία ακόμα φορά θέλω να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετικά επικοδομική συνεργασία και για την υποστήριξη που οδήγησε στην ε, έγκριση της συμφωνίας. Αυτό είναι σοβαρό επίτευγμα για όλα τα θεσμικά όργανα και μπορούμε από κοινού να πούμε ότι πράγματι όταν χρειάζεται μπορούμε να ε, συνεργαστούμε. Η συμφωνία αυτή έχει ενισχύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και έχει αυξήσει τη συλλογική μας ασφάλεια. Όταν συναντηθήκαμε τον Ιανουάριο κατά την ακρόαση μου σας είχα κάνει κάποιες υποσχέσεις. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα υποβάλω κάποιες ανακοινώσεις για την μετάδοση πληροφοριών και τα βασικά επιτεύγματα. Και τα δύο εγκρίθηκαν τον Ιούλιο. Έτσι λοιπόν τήρησα την υπόσχεσή μου. Ελπίζω να σας τα διαβάσατε γιατί φυσικά ζήτησα να σας ταλούν άμεσα. Η ανακοίνωση αφορά μια επισκόπηση όλων των μέσων ανταλλαγής πληροφοριών που υπάρχουν στην Ένωση ε, και στο θέμα της ασφάλειας και της διαχείριση τη μετανάστευση. Είναι μια μοναδική ε, μέθοδος αυτή γιατί στιγμή όλα αυτά τα μέσα ε, περιλαμβάνονται σε αυτό το, με αυτόν τον πολύ συνεκτικό και διαφανή τρόπο, έτσι ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι συστήματα υπάρχουν. Τα συστήματα όμως είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Υπάρχει όμως ένας πλήρης κατάλογός τους. Αυτό το πλαίσιο θα μας βοηθήσει να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πού χρειάζονται αυτά τα όργανα, πού δικαιολογούνται και αναφέρονται και κάποιες αρχές για τη χρήση τους. Και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει όταν θα τα επανεξετάζουμε αυτά. Η ανακοίνωση που ανέφερε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και επιτεύγματα για την καταπολέμηση τρομοκρατίας αναφέρει κάποιες σοβαρές δυσκολίες που υπάρχουν και αυτό είναι ένα από μακρού αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από κοινού τα έγγραφα αυτά μπορεί να αποτελέσουν μια σοβαρή βάση για την μελλοντική εξέλιξη της πολιτικής μας η Κομισιόν θα επιτρέψει, θα, σύντομα θα εγκρίνει ε, μια πρόταση για την απαγόρευση κάποιων χημικών ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν αυτοσχέδια εκρηκτικά και έτσι αυτό θα δυσκολέψει ακόμα τη, ε, την κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, τώρα με την άδειά σας θα αναφερθώ στις κάποιες πολιτικές ε, προτεραιότητες του φθινοπόρου. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο σας για την πολύ επικοδομητική προσέγγιση στο πακέτο PNR ε, εργαστήκαμε εντατικά το καλοκαίρι για να ολοκληρώσουμε μέχρι τον περασμένο μήνα τις διαδικασίες της Κομισιόν και με το ψήφισμά σα του Μαΐου σκοπός είναι να υπάρχει μια ανακοίνωση για την στρατηγική μας η οποία θα εγκριθεί από την Κομισιόν πριν το τέλος Σεπτεμβρίου. Ταυτόχρονα ως κομμάτι αυτού του πακέτου θα εγκρίνουμε προτάσεις εντολής για να, συν, για να συναυθούν τέτοιες συμφωνίες με την Αυστραλία, ΗΠΑ και τον Καναδά η ανακοίνωση για την εξωτερική στρατηγική PNR θα έχει κάποιες απαιτήσει και αρχές για μια τέτοια συμφωνία. Είναι σημαντικό οι αρχές αυτές να εγκριθούν πριν αρχίσουμε τι διαπραγματεύσει, για να υπάρχει λοιπόν ε, προστασία των δεδομένων και επίσης να υπάρχει μια ε, ξεκάθαρη εικόνα του ποια είναι τα προαπαιτούμενα. Βεβαίω πρέπει να υπάρχει κάποιο περιθώριο ε, λιγμών στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και τα ψηφίσματα, όμως οι αρχές που αναφέρονται είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτές που αναφέρατε εσεί στο ψήφισμά σας του Μαΐου. Τι. Τώρα, οι οδηγίες διαπραγμάτευσης θα αντικατοπτρίζουν αυτές τις αρχές. Φυσικά το Συμβούλιο θα πάρει την ε, τελική απόφαση, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να είναι συνεκτικές. Και χαίρομαι που αποδεχτήκατε ότι η συμφωνία με τις Ρωμαίες Πολιτείες και την Αυστραλία θα εξακολουθήσει να ισχύει στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προσωρινά όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων. Αυτό είναι απαραίτητο για να μην υπάρχουν κενά ασφαλείας και μια ε, και ένα ε, νομοθετικό κενό για τους αερομεταφορείς. Πάντως θέλω να συνεργαστώ πολύ στενά μαζί σας για να προωθηθεί το θέμα το ταχύτερο δυνατόν και θα κάνω μια ενημέρωση ε, για σας στη διάρκεια τη Συνόδου του στο Στρασβούργο την ερχόμενη εβδομάδα στις 21 του μηνός αφού ε, εγκρίνει τις, ε, προθέσεις, πρότασης της Κομισιόν. Όσον αφορά την, το, πακέ, της, το PNR της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία. Θα είναι ένα ευρωπαϊκό, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια μελέτη επιπτώσεων, όπως συνήθως κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που αναφέρεται και στο ψήφισμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πολύ σκληρά επίση για να προετοιμάσει μια ανακοίνωση για την εσωτερική στρατηγική ασφαλεία. Το Νοέμβριο θα βασίζεται ε, στα όσα αποφάσισε στην Ισπανική Προεδρία το Φεβρουάριο του Συμβούλιο Εσωτερικών και Δικαιοσύνη και θα συνάδει και με το πρόγραμμα αυτό και με το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη. Ε, θα ορίσει κάποιε βασικέ απειλέ, ε, οργανωμένο έγκλημα, έγκλημα στον κυβερνοχώρο, τρομοκρατία θεομηνίες ή ανθρωπογενείς φυσικές καταστροφές και με συγκεκριμένους στόχους για το πώς μπορούμε να είμαστε καλύτεροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτές τις απειλές. Βεβαίως πάντα ε, σεβόμενοι τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα προσωπικά δεδομένα και τις αρχές μας. Και στόχος είναι να βρούμε ε, πού μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί μόνο εφόσον υπάρχει ευρωπαϊκή υπεραξία και εκεί να συνεργαζόμαστε. Αυτή είναι η ατζέντα μας ε, και θα ήθελα να συμπεριλάβω και τις δικές σας προτάσεις και τις δικές σας ιδέες και παρακαλώ μην διστάσετε να τις υποβάλλετε σήμερα το απόγευμα. Μια μεγάλη προτεραιότητα για μένα κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου είναι το πακέτο για το άσυλο. Και είχα επαφές με εισηγητέ και σκιώδεις εισηγητέ της Επιτροπής σας από αυτού του θέματος. Ε, Κοινό σύστημα ασύλου είναι προτεραιότητα για μας να θεσπιστεί και ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει θέσει και χρονικό ορίζοντα το 2012. Το 2012 είναι κοντά μας και θα πρέπει τώρα να μεταφράσουμε αυτές τις πολιτικές δεσμεύσεις των κρατών μελών και των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων σε απτά και χειροπιαστά αποτελέσματα και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε ε, στη συνέχεια. Επίσης το θέμα επανεγκατάστασης. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας και ελπίζω το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να δείξουν ευελιξία για να μπορέσουμε το συντομότερο να συμφωνήσουμε. Δύο λόγια τώρα για την παιδική πορνογραφία και την καταπολέμηση ε, του εμπορίου ανθρώπων. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ για τις προτάσεις ε, της Επιτροπής σας και του Κοινοβουλίου. Έγινε μια ψηφοφορία ενδεικτική προσανατολιστική. Θα λάβουμε υπόψη την πρότασή σας και βεβαίως εξακολουθώ να υπολογίζω στην υποστήριξή σας για μια έκφαση συνεκτική και ισόρροπη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Είναι σύγχρονη δουλεία και δυστυχώ παρατηρείται και στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου. Γι' αυτό η καταπολέμηση του τράφικινγκ του εμπορίου ανθρώπων είναι πάρα πολύ μεγάλη προτεραιότητα για μένα και ελπίζω να βρεθεί λύση από τα τρία θεσμικά όργανα. Σχέδιο οδηγία κατά των επιθέσεων σε συστήματα πληροφοριών επίση θα εγκριθεί ε, αργότερα κατά τη διάρκεια του μηνό Σεπτεμβρίου, ελπίζω γρήγορα για να ενισχυθεί η νομοθεσία μα και ε, να οχυρωθούμε ε, στην προστασία μας από ε, εγκλήματα στο κυβέρνοχώρο. Βεβαίω ε, είμαι πρόθυμη να ακούσω τι ιδέες σα και το, για τη διαχείριση των συνόρων και τι μελλοντικέ ε, προτεραιότητε, Θα προτείνω ένα νέο μηχανισμό αξιολόγηση του Σέγγεν και ελπίζω να συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο, βέβαια πάντα σεβόμενοι το θεσμικό ρόλο του καθενό. Παρακολούθηση των όσων έχουν γίνει του τελευταίου μήνε και θα εγκρίνουμε ε, συστάσει για τη Μολδαβία, τη Ρωσία και την Ουκρανία για την απελευθέρωση των θεωρήσεων το συντομότερο και από τις χώρες αυτές. Προετοιμάζουμε επίσης διευκόλυνση θεωρήσεων ε, σε άλλα κράτη, Λευκορωσία, Αρμενία και Αζερβαϊτζάν που είναι στο σχήμα της γειτονίας. Ε, για ε, θεώρηση διαβατηρίων για άδεια σύντομη ε, παραμονή χώρες, από χώρε τη νότια όχθη Μεσογείου. Όπω βλέπετε, είναι πολύ μεγάλο το πρόγραμμά μα. Προσβλέπουμε σε εσά ω συνομοθέτε να συνεργαστούμε. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα. Υπολογίζω στη βοήθειά σα. Οι δικέ μου υπηρεσίε είναι πάντα στη διάθεσή σα. Τελειώνω. Πήρα το έγγραφό σα κυρία μου από τη Γαλλία Σήμερα το πρωί το διάβασα, διάβασα και στη Μοντ για πρώτη φορά υπέπεσε ε, στην αντίληψή μου. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικά αυτά που βλέπουμε. Χρειάζεται μελέτη και βεβαίως ε, εκτιμώντας και εξετάζοντας τι συνέβη στη Γαλλία θα τα λάβουμε και αυτά υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις σας. Παραμένω απολύτως στη διάθεσή σας, ρωτήστε με ό,τι θέλετε και θα κάνω ό,τι μπορώ. Και αν δεν μπορώ να σας απαντήσω, το συντομότερο θα σας φέρω την απάντηση. Thank you, Some members ε, ευχαριστώ. Ε, ζήτησαν το λόγο κάποιοι συνάδελφοι, αλλά καλό θα ήταν να ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές. Ε, τρία λεπτά έκαστος ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για το έργο σας μήνες πέρασαν από τότε που αναλάβατε και θέλω να σας ευχαριστήσω και για τον ενθουσιασμό σας και την ειλικρίνειά σας και την προθυμία συνεργασίας με την Επιτροπή μας. Είναι προφανέστατο από τον τρόπο που ε, συμπεριφέρεστε ότι διατελέσατε Ευρωβουλευτής και γνωρίζετε πολύ καλά ε, τι ε, θέλει το Κοινοβούλιο και πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο και πώς μπορείτε εσείς να συνεργαστείτε μαζί μας προς ε, το καλύτερο αμοιβαίο όφελος. Τούτου λεχθέντος, επιτρέψτε μου να αναφέρω μερικά σημεία τα οποία και εσεί αναφέρατε, ενώ κάποια άλλα δεν τα αναφέρετε. Να αρχίσω από τα όσα δεν είπατε. Μιλήσατε, μάλλον δεν μιλήσατε, για το αυξημένο τέλος που επιβάλλουν οι Ηνωμένε Πολιτείε στο ηλεκτρονικό σύστημα για έγκριση ε, ταξιδίων. Εγώ ό,τι ξέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έχει κοιτάξει αυτά από πέρυσι και τότε δεν είχε καταλήξει ότι αυτό ήταν επανεισαγωγή ουσιαστικά της θεώρησης με άλλο όνομα. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από την κίνηση αυτή και θεωρούμε ότι ένα σύστημα ελεύθερο θεώρησης διαβατηρίων θα πρέπει να είναι δωρεάν. Δηλαδή free στα αγγλικά σημαίνει ελεύθερο, σημαίνει και δωρεάν. Εδώ χρεώνουν 10 δολάρια. Για ένα σύστημα προώθηση των ταξιδίων το λένε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχονται και προσθέτουν και άλλα 4 δολάρια <laughs> για το διοικητικό, λέει, κόστος διεκπαιρέωσης ε, του φακέλου. Ε, ουσιαστικά, πρόκειται ε, περί επαναφοράς του στήματος θεώρησης διαβατηρίων με άλλο όνομα. Δεν το λένε Visa, το λένε κάτι άλλο. Ελπίζω και, και σας καλώ το συντομότερο και επιγόντως να το κοιτάξετε και να μας ε, ενημερώσετε για τις αποφάσεις που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και για τις προθέσεις της. Ε, περιμένω μεγάλη ενυπομονησία την απάντησή σας αυτό. Έρχομαι τώρα στο πακέτο για το άσυλο. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο το ζήτημα αυτό για σας να το αντιμετωπίσετε. Γνωρίζουμε ότι η θέση στο Συμβούλιο δεν είναι και η ευκολότερη. Υπάρχουν ε, προσκόμματα και εμπόδια που πρέπει να υπερβληθούν, αλλά με την ενέργεια και το, και το ενθουσιασμό που σας χαρακτηρίζουν, είμαι βέβαιος ότι θα ε, φέρετε σε αίσιο πέρα αυτή την προσπάθεια μέχρι το 2012 που θα είναι και η ώρα εφαρμογής του. Λείπουν ακόμα μερικά κομμάτια από αυτό το παζλ του πακέτου του ασύλου που θα θέλαμε να μελετήσετε και εσείς περισσότερο και ένα από αυτά είναι βέβαια το θέμα της ευθύνης και της, ε, του φόρτου και το κατά πόσο αυτό θα πρέπει να επιμερίζεται. Αλλά δεν υπάρχει νομοθετική πρόταση για την αλληλεγγύη. Έχουμε πιλωτικά προγράμματα και άλλες πρωτοβουλίες, αλλά κανένα νομοθετικό εργαλείο που να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο. Και θα θέλαμε και εμείς νομοθεσία και σε αυτό. Επίσης, στο ασυλό παραμένω, θα περιμέναμε συγκεκριμένα μέτρα που να στοχεύουν το θέμα της πρόσβασης στο άσυλο. Μιλήσατε για τα προγράμματα επαναγκατάστασης. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα. Αλλά επειδή προετοιμάζουμε ένα καλό πακέτο για το άσυλο, δεν δίνουμε καλές δυνατότητες εκείνους που θέλουν να κάνουν χρήση ε, αυτού του εργαλείου. Δεν τους δίνουμε ας πούμε νόμιμες οδούς και διάβλους για να ε, φτάσουν στο άσυλο στην Ευρώπη. Και επειδή δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία, βλέπουμε ακόμα καταστάσεις, ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη, όπου ο κόσμος προσπαθεί παράνομα και παράτημα να φτάνει στην Ευρώπη. Και μια τέτοια πρωτοβουλία με ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης που να λειτουργεί καλά στις τρίτες χώρες, θα υπάρχει και σωστή και θεμητή και τυπική πρόσβαση κανονικά στο άσυλο, όχι με αυτές τις μεθόδους. Βλέπω ότι ο πρόεδρος δυσανασχετεί και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ κύριε Μπούσουτιλ η κυρία Γκένς, η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Μάλμστρομ, σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή. Ε, ήταν ε, πάρα πολύ λεπτομερής. Βέβαια δεν μπήκε σε, σε επιμέρους θέματα γιατί ήταν τόσο ε, συνολική. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το TFTP, το Σύστημα Οικονομικού Εντοπισμού Τρομοκρατών. Ξέρετε ότι στο Κοινοβούλιο είπε ότι δεν ε, άρχισαν να ισχύουν με τον τρόπο που περιμέναμε ε, όλα τα στοιχεία της συμφωνίας από την 1η Αυγούστου. Μπορεί να είναι λανθασμένη αυτή η τύπωση που έχει δημιουργηθεί στο Κοινοβούλιο, αλλά θα πρέπει να μας ενημερώσετε, να απαντάτε στις ερωτήσεις μας, γιατί απευθύνονται και οι πολίτες σε εμά. Δηλαδή αυτή η βελτιωμένη συμφωνία πραγματικά λειτουργεί ε, καλά σε όλα τις τα ε, κεφάλαια, ας πούμε, όλα τα τμήματα. Και καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα πριν προχωρήσουμε στο PNR ή στην προστασία των δεδομένων για να μην ε, παραμένουν κρεμή ζητήματα που να μας προβληματίζουν. Σε αυτό το θέμα, στο TFTP, το σύστημα οικονομικού εντοπισμού των τρομοκρατών, θα ήθελα κατά τη διάρκεια του μηνός να το ξανασυζητήσουμε. Θα ήταν χρήσιμο για όλους τους ενεχομένους ε, θα ήθελα να σας κάνω ξανά όμως κάποιες ερωτήσεις. Τα κριτήρια, όχι μόνο για την επιλογή στη Europol, τους υπαλλήλους δηλαδή πώς επιλέγονται αυτοί που ε, ελέγχουν αυτά τα στοιχεία, αλλά τι γίνεται και με τους υπαλλήλους της εφορίας. Το ποιοι είναι αυτοί, δεν ρωτάμε εμεί τα ονόματα, αλλά εννοούμε τι προσόντα και δεξιότητες και γνώσεις έχουν αυτοί οι άνθρωποι που διαχειρίζονται αυτά τα στοιχεία. και στην Αμερικανική εφορία. Δεν είναι τεχνικό αυτό το έργο για το καθήκον, γιατί είναι θέσεις ευθύνη και θα πρέπει να καταλαβαίνουν και την πολιτική διάσταση της δουλειά τους, όχι να πατάνε κάποια κουμπάκια σε κάποιους υπολογιστέ και μόνο. Κάτι άλλο. Ποιος αποφασίζει σε τελική ανάλυση ποια πακέτα δεδομένων ε, διαβιβάζονται και πώς γίνεται η συνεργασία μεταξύ εφορίας, ευρωπόλ, τραπεζών και τα λοιπά και τις εταιρείες που τα έχει αναλάβει όλα αυτά. Πώς γίνεται η επικοινωνία. Είναι ασφαλής. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα μπορέσετε να απαντήσετε σε όλα αυτά τα θέματα, αλλά καταλαβαίνετε πόσα ερωτηματικά μας έχουν ε, ακόμα Τώρα, για την διατήρηση, αποθήκευση και κράτηση αυτών των στοιχείων και των προσωπικών δεδομένων. Εσείς το βλέπετε αυτό κυρίως ως πρόβλημα εφαρμογής στα κράτη-μέλη. Αυτό δεν λειτουργήσε σωστά. Ή μήπω σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να κάνουμε αλλαγές προς την κατεύθυνση αυτή και να διευκολύνουμε τα κράτη-μέλη για να εφαρμόζουν αυτή την οδηγία. Ή απλώς είναι ένα θέμα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Ένα τελευταίο για την παιδική πορνογραφία. Γνωρίζετε όπως και εγώ ότι συχνά στη συζήτηση κυριαρχεί το θέμα ε, της ε, διαγραφής ε, και της πραγής από τους υπολογιστές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και πολλά άλλα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ εντατικά, θέματα που περιλαμβάνονται στην οδηγία. Και ένα τελευταίο για το πακέτο του ασύλου. Ένα λιγότερο ίσως σημαντικό. Ο κύριος τι είπε ότι είναι δύσκολο να συμφωνεί στο Συμβούλιο γιατί υπάρχουν προβλήματα και προσκόμματα. Αλλά Εμένα με ανησυχεί ε, που αυξάνεται και ο αριθμό των συμφωνιών για τις λεγόμενες ασφαλείς χώρες προέλευσης ή διέλευσης. Εσείς πώς το αξιολογείτε αυτό, γιατί όλο και περισσότερο προβληματικά κράτη χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται στην κατηγορία των ασφαλών. Ε, ευχαριστώ. Για την ομάδα των φιλελευθέρων, κύριε Έλπε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ καλωσορίζω την κυρία Μάλστρομ, την Επίτροπο. Θέλω να πω ότι πράγματι τα... η θεματολογία της υπήρξε από την αρχή φιλόδοξη και εξακολουθεί να είναι φιλόδοξη. Είμαι ιδιαίτερος ευγνώμων που ήρθατε στην Επιτροπή μας για να μας ενημερώσετε για το... την κατάσταση στην οποία βρίσκονται όλα αυτά τα θέματα και το, την εξέλιξη της δουλειάς σας. Θέλω να σας θέσω ε, δύο θέματα. Πρώτον, το TFTP και τον διορισμό αυτών οι οποίοι θα εργαστούν εκεί. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες της Κομισιόν για ολόκληρη αυτή τη διαδικασία, για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της δουλειάς και αυτών οι οποίοι θα απασχολούνται εκεί. Και παρότι το καταλαβαίνω πρέπει να υπογραμμίσω ότι όλη μου τη ζωή η εμπειρία μου είναι ότι τα παιδιά είναι για τους έντιμους, όχι για τους ε, εγκληματίες. Εμείς οι έντιμοι δεν θα ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, οι άλλοι όλοι θα ξέρουν αυτό, περί αυτού να είστε βέβαιοι. Έχουν δικού του τρόπους να μάθουν αυτά που θέλουν. Στην ουσία είναι αδύνατον τα ονόματα αυτά να παραμείνουν κρυφά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ενδιαφέρει εμάς δεν είναι το όνομα αυτό καθεαυτό. Μάλλον η συνολική διαδικασία βάσει της οποίας θα γίνονται οι αναφορές προς εμάς. Είναι σημαντικό συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε. Πρέπει να ενημερωνόμαστε για το αν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Γιατί αυτό είναι κάτι που αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι αναφορές προς το Κοινοβούλιο θα γίνονται σωστά και δεν μπορούμε ξεκινώντας να πούμε ότι δεν ε, εμπιστευόμαστε τα άτομα αυτά ή ότι αυτά θα καλύπτουν ε, τις ατασταλίες, αλλά βεβαίως ε, ως κοινοβουλευτικός κανείς πρέπει να είναι καχύποπτος, έτσι πρέπει να είναι. Αλλά αν με ρωτήσετε, αυτό αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για να έρθει κανείς στο θέμα της διπλής αυτής ε, διαδικασίας, της δυνατότητας ε, απο, ε, απο, στοιχείων από προσωπικών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η πολιτική μου ομάδα θέλει να παραμείνει εντός του πακέτου και όχι στο πλαίσιο της βαθμίας προσέγγισης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άλλες απόψεις στο Συμβούλιο. Θεωρώ ότι μπορούμε να ακούσουμε και άλλες προτάσεις για το πώς εμείς οι ευρωβουλευτές μπορούμε να βοηθήσουμε να απεμπλακούν οι συζητήσεις και η συζήτηση, η λήψη απόφαση του Συμβούλιο. Και συμφωνώ με τον Σάιμον που αναφέρθηκε στην ε, κατανομή των ευθυνών και στην αλληλεγγύη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπωσδήποτε δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση το βάρος βρίσκεται περισσότερο σε με κάποιες χώρες και όχι σε όλες. Μιλάμε για σύνορα Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης. Επί του άλλου θέματος μία μόνο παρατήρηση. Και για την ε, παιδική πορνογραφία, τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας και όλα αυτά τα θέματα. Πάντοτε ήμουν και θα εξακολουθήσω να είμαι αρνητική σε νομοθεσία, καχύποπτη απέναντι σε νομοθεσία που προσπαθεί να ε, περιορίσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί ο υπόλοιπος κόσμος δεν κινείται έτσι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πάντα υπάρχει μια τάση να επιβάλλουμε αυστηρότερους κανόνες στους εαυτούς μας, παρότι ο υπόλοιπος κόσμος απολαμβάνει άλλες καταστάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλμπρεχτ για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω επιπλέον ερωτήσεις. Μια σύντομη πρώτα προς την κυρία Μάρσον. Η ολοκλήρωση του ΣΥΣ 2 έχει νόημα, είναι ρεαλιστικό, όλο αυτά μας τρώει αυτή η υπόθεση. Το σύστημα προφόρηση Σέγγεν δηλαδή είναι αυτό. Ε, μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιες εναλλακτικέ λύσεις ε, υπόθεση. Και μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπε και η κυρία Βέμπερ για το σύστημα οικονομικού εντοπισμού των τρομοκρατών. FTP. Αναρωτιέμαι κι εγώ για αυτά τα θέματα και για ένα ζήτημα αμοιβαιότητας για την αμοιβαία νομική συνδρομή Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Τι γίνεται με άρθρο 4 της ατομικής μεταφοράς στοιχείων, μεμονωμένης μεταφοράς τραπεζικών στοιχείων. Οι ΙΠΑ εφαρμόζουν αυτό το άρθρο όταν πρόκειται για τραπεζικά στοιχεία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά για ε, υποθέσεις που εκκρεμούν στη δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Και αυτό που είπε η κυρία Σίπελ για την αποθήκευση των στοιχείων. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα γίνει μια αναθεώρηση και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλήσετε για αυτή την ανακοίνωση για το πώς έχουν τα μέτρα ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό άλλωστε και ως ε, βουλευτές εμείς το ζητούμε πάγια. Αλλά θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση πραγματικά προς εσάς κυρία Μάστομα ότι θα πρέπει να παρακολουθείτε και τις διαδικασίες που τρέχουν στη δικαιοσύνη. Από τότε που εγκρίναμε την οδηγία υπάρχουν πολλές υποθέσεις στα εθνικά δικαστήρια και μία φτάνει πλέον και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχει έρθει λοιπόν πλέον ο χρόνος να αναθεωρήσουμε όλο αυτό το θέμα της υποχρέωσης αποθήκευσης αυτών και των τηλεφωνιών στοιχείων και των τηλεπικοινωνιών και πώς ε, ρυθμίζεται και αυτά τα θέματα με τις εθνικές κυβερνήσεις. Και ένα τελευταίο σχόλιο μάλλον, δεν είναι ερώτηση. Όταν έχουμε ποινικέ διώξεις, είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει χάσμα και διαφορά άμεσα στο δικό σας χαρτοφυλάκιο και εκείνο της κυρίας Ρέντινγκ. Γιατί, ας πούμε, συνεργαζόμαστε για τα προσωπικά στοιχεία των επιβατών, αυτό το PNR. Και μετά είμαι εγώ εισηγητής για τη γενική προστασία των δεδομένων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπα, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε σε ποιον απευθυνόμαστε και να είναι συνεκτική η θέση και ενιαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το λέω από τώρα πριν αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Όπως επίσης και το θέμα ε, των, ε, της κακοποίησης παιδιών, ε, τις ποινικέ κυρώσεις ας πούμε. Ποια είναι τα δικονομικά δικαιώματα ας πούμε. Και πώς θα εναρμονίσουμε τις ποινικέ κοινώσεις σε τέτοιες διαδικασίες ποινικού δικαίου, γιατί πολλές χώρες ανησυχούν. και χρειάζεται εναρμόνιση, πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Thank you. For Mr. Tavares. για την Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με την TFTP για να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Η μυστικό της που διέπει την επιλογή των ε, Ευρωπαίων ε, στην Ουάσιγκτον δεν αφορά, δεν έχει την, την συμφωνία ή την ε, διαπραγμάτευση που θα γίνει στο μέλλον. Δεν είναι αυτό που θέλαμε, ούτε αυτό που μας υποσχέθηκαν και επίσης επί του TFTP. Τι έγινε τον Ιούλιο και γιατί στις αρχές Ιουλίου η υπογραμματεία ε, ε, κατά της τρομοκρατίας από ε, ε, τις ΟΠΑ μας είπαν ότι τα SWIFT data ήδη ε, συλλαμβάνουν ε, τρομοκράτες όταν δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η μεταφορά δεδομένων γιατί η, σύμφωνα με τη συμφωνία αυτά θα έπρεπε να αρχίσουν μετά την 1η Αυγούστου. Άρα ε, θα ήθελα να μάθω ε, αν έγιναν τέτοιες ε, αποστολές δεδομένων ή όχι. Και επίσης συμφωνώ με αυτό που είπε ο Γιαννάπερς για τις μεταφορά τραπεζικών δεδομένων από τις Ηνωμένε Πολιτείε προς την Ευρώπη και το σχετικό άρθρο της Συνθήκης Αμοιβές Δικαστικής Συνθρομής. Τώρα, έχω, είμαι πολύ περίεργος για την ανακοίνωση που προετοιμάζει η Κομισιόν για την εσωτερική ασφάλεια και θεωρώ ότι είναι πολύ ε, ενδιαφέρον που υπάρχουν φυσικές καταστροφές σε αυτή την ανακοίνωση. Ελπίζω να υπάρχει μια διευκρίνηση ας πούμε, στη χρήση συγκεντρωμένων πόρων, σε σχέση, συγκέντρωσης πόρων για τις φυσικές καταστροφές, ιδίως διαμεθοριακές ε, φυσικές καταστροφές όπως οι δασικές πυρκαγιές. Υπήρξε ας πούμε ένα θέμα φέρει στο καλοκαίρι. Η χώρα μου δεν χρησιμοποίησε ε, αυτά που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στο, στην πυρόσβεση και πολλοί μου λένε ότι αυτό συνέβη διότι αφού να βλώσει κανείς τα αεροσκάφη, το κράτος μέλος πρέπει να πληρώσει το μισό ε, κόστος ε, εντός 190 ημερών και για χώρες που πλήττονται από αυτή την κρίση ίσως αυτό να γίνεται να είναι δύσκολο και να μην υπάρχει αυτή η οικονομική δυνατότητα. Οπότε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε τις δασιοικές πυρκαγιές με τα μέσα που θεωρούσαμε ότι θα είχαμε στη διάθεσή μας. Επίσης αναφερθήκαμε επανειλημμένως στο... Ε, είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν προχωρήσουμε θα υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον και κυρίως θα χαθεί αυτή η ε, καλή αρχή που έχει γίνει για την επανεγκατάσταση και την υποδοχή των αναμεκαταστηθέντων ε, προσφύγων. Υπάρχει αυτή η έκθεση όπου το Συμβούλιο είχε θέσει ε, μια κόκκινη γραμμή σε σχέση με δημοσιονομικά θέματα και συνεχώς λέω ότι αυτό δεν είναι ένα δημοσιονομικό θέμα. Είναι ένα θέμα ε, περιφερειακής πολιτικής και άρα απόφαση εξωτερική ε, ε, που σχετίζεται με εξωτερική πολιτική. Επίσης, όσον αφορά την πολιτική αποκατάσταση συστημάτων των βασανιστήριων, την υποστηρίζαμε αυτή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα ε, ξαφνικά μοιάζει ότι σιγά σιγά ε, σταματά η στήριξη των τέτοιων κέντρων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως το 20-30% των θυμάτων που υπάρχουν είναι θέματα, ε, θύματα βασανιστήριων, έχουν μετέπειτα στη ζωή τους προβλήματα και ο λόγος που σταματά αυτή η υποστήριξη είναι ότι ήταν μια πρωτοβουλία ε, των εξωτερικών σχέσεων. Πιστεύω ότι πρέπει να καλύψουμε αυτό το κενό στον τομέα της εσωτερικής πολιτικής και να δημιουργηθούν νέα χρηματοδοτικά μέσα για τα κέντρα αποκατάστασης θυμάτων βασανιστήριων. Ίσως ε, στην ε, συζήτηση για τον προπολογισμό να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από την ομάδα των συντηρητικών ε, και μεταρρυθμιστών, κανείς δεν θέλει το λόγο. Από τους μία εγγεγραμμένου, ο κύριος Μπρόνς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι από τους μη εγγεγραμμένους, αλλά δεν μιλώ εξ ονόματός τους, μιλώ για τον εαυτό μου. Η Επίτροπος μίλησε για μια ταχεία διαδικασία για ειδικευμένου ε, εργάτες, εργαζομένους. Ακούσατε την περασμένη εβδομάδα ε, στο κοινοβούλιο την ομιλία που έλεγε ότι 53% ήταν ο πρόεδρος του Μαλή που είχε μιλήσει και είπε ότι το 53% των πτυχιούχων ε, της χώρας το εργάζονται στο εξωτερικό και ε, τους παίρνουμε υγειονομικό προσωπικό που είναι πάρα πολύ καλά μορφωμένο και το στερούνται αυτές χώρες, χώρες όπως το Μαλή. θα πρέπει δηλαδή να εξαφανιστούν και να πεθάνουν γιατί δεν μπορούν οι ίδιες μας οι χώρες να ε, εκπαιδεύσουν το προσωπικό του ε, σε άλλες ειδικότητε. Αυτό μπορεί να μην έχει τόσο τραγικές συνέπειες, αλλά μπορεί ε, να καταδικάσει χώρες όπως το Μαλή να παραμένουν φτωχές σε ΣΑΗ. Μεγάλο σεβασμό έδειξε στον πρόεδρο του Μαλή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφήνοντά τον να μιλήσει. Θα είχε δείξει μεγαλύτερο σεβασμό το Κοινοβούλιο να άκουγε για αυτά που έλεγε ο άνθρωπο. Υπάρχουν πολλοί που φεύγουν από χώρες ασφαλείς, ε, τις παρακάμπτουν και ε, ζητούν άσυλο. Ε, και ορισμένοι όμως είναι γνήσιοι τούντες άσυλο, υποφέρουν γιατί έρχονται από χώρες που κινδυνεύουν. Αυτή είναι η λογική του ασύλου. Δεν θα πρέπει να τη δώσουμε την πραγματική της διάσταση και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ας διευρύνουμε λοιπόν ε, την εικόνα με τα μέλη που ενδιαφέρονται. Η κυρία Ιντβελτ. Μήπως θέλετε να απαντήσετε πρώτα, κύριε Επίτροπε. Βεβαίω. Λοιπόν, να κάνουμε μια πρώτη σειρά, να δώσουμε μια πρώτη σειρά απαντήσεων και μετά να πάρουν το λόγο τα υπόλοιπα μέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με αυτόν τον τρόπο θα απαντήσω ίσως κάποια ερωτήματα που και θα μην ε, επανέλθουν. Κύριε Μπουζούτη, κύριε για το έστωφι. Ναι, πράγματι έχω θέσει το θέμα στις Αμερικανικές Αρχές και έχουμε ασχοληθεί. Είναι ενοχλητικό. Λάβαμε πολλά παραδείγματα, ε, πολλά ε, παράπονα από επιπλέον από πολίτε, Ναι, αυτό το επιπλέον κόστος το έχουμε θέσει στου Αμερικανού και έχω ζητήσει από τη Βελγική Προεδρία να το θέσει στο επόμενο Συμβούλιο Τζάι για να δούμε πώ θα αντιδράσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης συνεργαζόμαστε χωρίς να προκαταλαμβάνω φυσικά τα αποτελέσματα αλλά κάνουμε ε, μια μελέτη επιπτώσεων τη Ευρωπαϊκή Πληροφορίας. Βεβαίω ενοχλεί αυτό τους Ευρωπαίους πολίτες για το πακέτο του ασύλου. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας αλλά χρειάζομαι και τη βοήθειά σα. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εισηγητών για να προχωρήσω στον τομέα αυτό. Ε, κάποιες από τις προτάσεις είναι απλούστερες από άλλες, αλλά εν πάση περιπτώσει όλες έχουν τις δυσκολίες τους. Θα συζητηθεί αύριο στην διάσκεψη των Υπουργών που οργανώνει η Βελγική Προεδρία και θα υπάρξει και αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέματα ασύλου, όχι διατρέχοντας τις προτάσεις ε, μια προς μία, αλλά το θέμα γενικότερα και ελπίζω ότι αυτή η διάσκεψη θα μπορέσει να ε, μας δώσει μια γενική εικόνα ε, της διάθεσης και μετά θα έρθω σε εσά να συζητήσουμε στις στρατηγικές πρόοδου. Η ελεγγύη είναι σημαντική. Πραγματικά εν μέρει αυτό φαίνεται στο πακέτο του ασύλου, αλλά του χρόνου η Κομισιόν θα υποβάλει μια ανακοίνωση και μια πρόταση για την ενδοευρωπαϊκή αλληλεγγύη με βάση τα πιλωτικά προγράμματα και άλλες ιδέες που ήδη υπάρχουν. Ήδη συγκεντρώνουμε ιδέες και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω και τις δικές σας ιδέες. Η κυρία Σίπελ και πολλοί άλλοι ρώτησαν για το τι πρόγραμμα TFTP. Ε, η συμφωνία έχει τεθεί ενισχύει από την πρώτη Ογδόου. Φυσικά δεν κατέστη δυνατόν από την πρώτη μέρα να υπάρχει εκεί ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν. Προχωρήσαμε όμως το ταχύτερο δυνατόν και υπάρχουν προσωρινά εργαζόμενοι Ευρωπαίοι πολίτες στη Ουάσιγκτον από το τέλος Αυγούστου. Υπάρχει Ευρωπαίος πολίτης που έχει σχετική εμπειρία που έχει ε, έγκριση των Αμερικανικών αρχών και κάνει την καθημερινή παρακολούθηση όπως προβλέπει η συμφωνία. Ε, ενημέρωσα τον εισηγητή γιατί αυτό έγινε εν μέσω καλοκαιριού, ήταν ε, δύσκολο να έρθουμε σε επαφή με όλους σας. Φυσικά δημοσιεύσαμε τη θέση, το κάναμε έγκαιρα. Η προθεσμία ε, λίγη την Τετάρτη ε, υποβολής αιτήσεων και όταν θα έχουμε τον κατάλογο θα βρω τρόπους να συζητήσω μαζί σας για τα κριτήρια. Φυσικά η θέση είναι θέση τεχνική, όχι πολιτική. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάποιον που θα πάει να δίνει συνεντευξείς. Είναι ένας άνθρωπος που θα πηγαίνει καθημερινά για να παρακολουθεί τη δουλειά, όλες τις ε, ε, επιταγές, ε, είναι μια τεχνική δουλειά, όλα τα εμβάσματα κλπ. Πρέπει λοιπόν το άτομο αυτό να έχει κάποια εμπειρία στον τομέα και βεβαίως πρέπει να εγκριθεί ο διορισμός και από τους Αμερικανούς. Το Σεπτέμβριο έχει προβλεφθεί μια κεκλεισμένο των θυρών συνάντηση όπου μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιλογής και τα κριτήρια που απαιτούνται. Έχω ενημερώσει επίσης όλους τους συντονιστές για αυτά τα οποία σας είπα. Φυσικά θα υπάρχει μια ομάδα επανεξέτασης που θα μελετά το θέμα. Άρα ε, ο άνθρωπος αυτός δεν θα αναφέρεται καθημερινά στην Κομισιόν, θα είμαστε όμως σε επαφή μαζί του και η, η, η συμφωνία αναφέρει ότι έξι μήνες μετά την θέση ενισχύτη της ε, συμφωνίας θα υπάρξει μια ομάδα μελέτης η οποία φυσικά θα έρθει σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Οι βελγικές και οι ολλανδικές αρχές από... έχουν προσφέρει τις δικές τους αρχές προστασίας δεδομένων, μέλη για να συμμετάσχουν σε αυτή την ομάδα ελέγχου. Ήδη έχουν ε, ξεκινήσει προετοιμασία για το ευρωπαϊκό TFTP, αυτό το ρώτησαν κάποια, άλλα μέλη, μετά τις προθεσμίες και τα χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στη συμφωνία και ελπίζω ότι θα μπορέσω να σας ε, υποβάλω ε, κάποιες από αυτές τις ιδέες μετά τη μελέτη επιπτώσεων και θα σας ενημερώνω και για όλα αυτά τα ζητήματα και όλες τις εξελίξεις. Επίσης για το TFTP, κύριε Ταβάρες, ο Υφυπουργός κύριος Λέβη νομίζω αναφέρθηκε στην ε, σύλληψη, ε, στο σταμάτημα κάποια σχεδιαζόμενης τρομοκρατικής επίθεσης στην Ορβηγία το καλοκαίρι. Αυτό βασιζόταν σε περασμένα στοιχεία, γιατί υπήρχε όπως είπατε μια ε, διακοπή μεταφοράς των δεδομένων από την εποχή που εσείς το Μάιο καταψηφίσατε μέχρι τον Αύγουστο και επίση, οι δύο, δύο, τις δύο, δυόμιση εβδομάδες του Αυγούστου δεν υπήρχε καμία μεταφορά δεδομένων. Άρα τα δεδομένα που οδήγησαν ε, στην αντιμετώπιση αυτής της συνωμοσία τη Νορβηγίας στηριζόταν σε ε, μεταφορά δεδομένων παλαιότερα. Ελπίζω κύριε Πρόεδρε να απάντησα σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν το TFTP. Ε, με τα χαρά θα επανέλθω για να μπω σε λεπτομέρειες και να δώσω και γραπτές απαντήσεις αν υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε γιατί πραγματικά προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη διαφάνεια. Για την παιδική πορνογραφία, ναι, θα γίνει συζήτηση το Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Αυτό προβλέπεται Γνωρίζω ότι υπάρχει ευρία στήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν γίνει όμως ερωτήσεις για την πρόταση της Κομισιόν για το κλείσιμο στην πηγή, πάντα το καλύτερο, αλλά επίσης ε, επιπλέον ε, και το μπλοκάρισμα των σελίδων ε, παιδικής πορνογραφίας φυσικά με πάρα πολύ αυστηρές διατάξεις και υποέλεγχον. Αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι οι εταίροι, οι εμπλεκόμενοι να διαπραγματευτούν. Τώρα για την παρακράτηση στοιχείων το συζητάμε ε, για, ε, δουλεύουμε να κάνουμε την, την αξιολόγηση. Έχουμε σοβαρά προβλήματα τα κράτη-μέλη. Δεν στέλνουν τις απαντήσεις και τις απόψεις τους. Γιατί όποια και είναι η απόψή σα για την οδηγία και ξέρω τις απόψεις πολλών από τα μέλη, η σωστή αξιολόγηση πρέπει να στηριχθεί για το, με το βάση του πώς έχει χρησιμοποιηθεί, ε, έχει προσφέρει υπηρεσίες, για ποιο λόγο και τα κράτη-μέλη ε, δεν μας απήντησαν γρήγορα. Το έχω πενθυμίσει επανελειμμένος. Γι' αυτό η αξιολόγηση έχει κάπως καθυστερήσει. Ελπίζω όμως ότι οι απαντήσεις θα έρθουν στις επόμενες εβδομάδες και θα μπορέσω να τις συζητήσω και με εσά και με τον εισηγητή. Δεν ξέρω αν υπάρχει ήδη εισηγητής επ' αυτού. Πακέτο ασύλου. Η, προμοθε... η προθεσμία είναι το 2012. Τότε πρέπει να υπάρχουν όλα. Έχουμε πει και με την ε, Βελγική Προεδρία έχουμε εντοπίσει κάποια εύκολα θέματα. Το Eurodac ας πούμε, τα προσόντα και η μακράς διαρκείας παραμονή έχει γίνει πρόοδος. Επί του Δουβλίνου έχουν, υπάρχουν κάποια δύσκολα ζητήματα, κυρίως ε, όσον αφορά έναν πιθανό μηχανισμό αναστολής, όπου υπάρχει ελάχιστη θα έλεγα, ε, πάρα πολύ μικρή στήριξη στο Συμβούλιο για τις ε, προθέσεις κομισιών, δύο-τρία μέλη μόνο μας υποστηρίζουν. Επίσης υπάρχουν και, άλλες, άλλα ζητήματα, οι διαδικασίες, οι, οδηγίες διαδικασίας και υποδοχής είναι πιο δύσκολε. Ελπίζω όμω ότι και αυτέ θα έχουν, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2012 ε, όπως έχει ομόφωνα αποφασίσει το Συμβούλιο. Τα δύσκολα είναι κάποια οριζόντια θέματα και ελπίζουμε ότι προχωρώντας και διεκπεραιώνοντα κάποια από αυτά ε, τώρα μπορούμε να, να ξεπεράσουμε κάποιε δυσκολίε. Όμω πραγματικά χρειάζομαι την υποστήριξή σα γιατί υπάρχει μεγάλη αντίδραση στο Συμβούλιο. Επί το ΣΥΣ2, κυρία ναι, τηρήσαμε το χρονοδιάγραμμα όπως σας είχα πει στο Συμβούλιο. Υπάρχει, ε, προετοιμαζόμαστε για το δεύτερη ημερομηνία ε, και ελπίζω, ε, ε υπόσχομαι ότι το τέταρτο πέμπτο Συμβούλιο θα υπάρχει σχέδιο και προπολογισμό που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο αλλά και σε εσά για να κάνετε και εσείς τις εκτιμήσεις σας. Είμαστε όμως ε, στο, στον καλό δρόμο, παρακολουθούμε το χρονοδιάγραμμα. Για, όσον αφορά τα δεδομένα σας απίτσα και εσείς και άλλοι έθεσαν το θέμα της ε, αλληλεπικάλυψης των δικών μου αρμοδιοτήτων με τον αρμοδιότητα της κυρίας Ρέντινγκ. Αυτό είναι λίγο φυσιολογικό. Ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο διαιρέθηκε στα δύο, αλλά έχουμε καλή και στενή συνεργασία επί όλων αυτών των θεμάτων και είμαι βέβαιος ότι και εκ μέρους μπορώ να πω ότι αν θέλετε να μας καλέσετε και τις δύο στην Επιτροπή να συζητήσουμε κάποια θέματα, σαφώς μπορούμε να το κάνουμε. Όσον αφορά την εσωτερική στρατηγική ασφάλειας, η, κύριε Ταβάρης, μία από τις ε, απειλές εδώ είναι ο τρόπος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανθρωπογενείς ή μη ανθρωπογενείς ε, φυσικές καταστροφές, τον νέα ρήτρα δηλαδή που προβλέπει συνθήκη. Δεν θα υπάρχουν συγκεκριμένες δημοσιονομικές προτάσεις από αυτού φυσικά, αλλά ένας τρόπος για το πώς θα ε, χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας για την αξιολόγηση κινδύνου και τον τρόπο καλύτερη δυνατή χρήση. Όσον αφορά το θέμα της αποκατάστασης θυμάτων ε, ε, βασανιστήριων, σας ευχαριστώ που, δεν, που το θέσατε, δεν το γνώρισα, θα το συζητήσω με την κυρία Άστον, με τον κύριο Μπρόντσο. Ε, το θέμα της, των, της μετακίνησης υπαλλήλων εταιριών αφορά κάποιες λίγες πολυεθνικές, δεν αφορά νοσηλευτικό προσωπικό γιατρούς, κυρίως αφορά μηχανικούς και ειδικούς υπολογιστές κυρίω 60.000 είναι αρκετοί, αλλά είναι οι εμπειρογνώμονε αυτών των επιχειρήσεων. Και εν γέννη θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να μετακινούνται οι άνθρωποι, να παίρνουν εμπειρίε και να επιστρέφουν στις χώρες τους με κάποιες νέες εμπειρίες και νέα χρήματα. Υπάρχει λοιπόν ένας κύκλος μετανάστευσης για τους αιτούντες άσυλο. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει ατομική αξιολόγηση. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν υπογράψει σύμβαση της Γενέβης και όλοι οι αιτούντες άσυλο από όποιαν προέρχονται και υπό οποιασδήποτε συνθήκες έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεως ασύλου και ατομικής αξιολόγησης. Η Κομισιόν δεν έχει σκοπό να κάνει τίποτα για να περιορίσει αυτή τη δυνατότητα της ατομικής ε, αίτησης ασύλου. Ευχαριστώ. Εγώ σα ευχαριστώ. Τώρα ο δεύτερος γύρος, η κυρία Ινετφέλτ, στα αγγλικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Με χαρά σα βλέπουμε πάντα ενώπιον μα Δύο θέματα θα ήθελα εγώ να θίξω. Πρώτον, το θέμα των Ρωμά. Ανέφερε και η κυρία Βερζιά ε, τις εξελίξεις. Μάθαμε το Σαββατοκύριακο τα νέα διέρευσαν κάποια έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η γαλλική κυβέρνηση εσκεμμένα ε, στόχευε καταβλισμού στον Ρωμά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα με τους Ρωμά. Την περασμένη εβδομάδα το Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τη στρατηγική που αρμόζει. Ωστόσο, η συλλογική ε, απέλαση ανθρώπων βάσει εθνοτικά κριτήρια είναι πάρα πολύ βαρύ ζήτημα. Και θα παρακαλούσα και εσάς και τη συνάδελφό σας κυρία Ρέντι ε, η οποία ήταν ελαλίστατη για αυτό το θέμα να, ε, και σε υψηλούς τόνους, να κάνει τις δικές της έρευνες και να μην επαφίεστε σε αυτά που λέει η γαλλική κυβέρνηση αν υπήρχαν αιτιάσει για παράνομα καρτέλ ή παράνομε κρατικέ ενισχύσει, θα κάνετε κι εσεί ξεχωριστή έρευνα και δεν θα πιστεύατε το λόγο της προσκοπικής τιμής που δίνει μια κυβέρνηση. Τώρα για τους καταλόγους με τα ονόματα των επιβατών, το PNR, ελπίζω την άλλη εβδομάδα να εγκριθεί αυτό. Ξέρω ότι προσωπικά είστε πάρα πολύ ε, προσιλωμένοι στις συστάσεις του Κοινοβουλίου και θέλετε να τις ακολουθήσετε. Ελπίζω το κολέγιο, έτσι, το συνολικό σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σας ακολουθήσει τη σοφία σας. Ξέρετε, εγώ θέλω να θυμίζω πάντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εμείς είμαστε με το χέρι στο κουμπί ακόμα γιατί πρέπει να ψηφίσουμε τις συμφωνίες αυτές και υπάρχει και προθεσμία. Και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το εγκρίνει και να τα αποκριθεί την άλλη εβδομάδα για να υπάρξει επιτέλους κοινή θέση μεταξύ ε, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί το σφάλμα που κάναμε με το SWIFT που εμφανιστήκαμε διχασμένοι Ευρωπαίοι να μην επαναληφθεί. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα εδώ να σας ρωτήσω είναι το εξή. Είδαμε αλλού το πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων διαβατήριων, αλλά βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα για να πιέζουν κυβερνήσει κρατών μελών, που θέλουν ας πούμε, να εξαιρεθούν από, τη, από την ε, θεώρηση ή να παραμείνουν ε, ελεύθερα θεώρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας δώσει μια επισκόπηση των διμερών συμφωνιών ή ε, διαπραγματεύσεων για την κατάργηση θεώρησης και σε ποιο βαθμό παίζει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ρόλο το PNR. Γνωρίζουμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι όλες οι κυβερνήσεις πάρα πολύ ειλικρινείς και δεν το συζητούν ανοιχτά, αλλά θα θέλαμε να έχουμε μια ιδέα παραπάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο Κοέγιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επίτροπο, κυρία Μάστρομ, ε, που ήρθε και για την ομιλία της. Και θα χαιρόμουν πάρα πολύ να μας δίνατε και ένα αντίγραφο της δήλωσής σας, ένα κείμενο, γιατί βρήθη σημαντικών στοιχείων. I welcome your... ε, σας ε, καλωσορίζω και χαίρομαι για αυτά τα θετικά που είπατε και τα αισιόδοξα για το ΣΥΣ. Έχετε καθόλου κανένα χρονοδιάγραμμα, έστω και προσωρινό, ε, για να δούμε πώς θα πιέσουμε τις εξέλιξεις. Δεν άκουσα να είπατε τίποτα για το ΒΙΣ, όχι για το ΣΥΣ. Ε, έχετε τίποτα νέα να μοιραστείτε μαζί μας. Επίσης, χάρηκα και αυτό που είπατε για το σύστημα ε, αξιολόγησης του Σέγγεν. Είπατε με τρόπο πάρα πολύ εύστοχο ότι το Κοινοβούλιο και διπλωματικό θα ασχοληθεί με το θέμα. Τι εννοείτε. Πότε θα το κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Είναι στη διαδικασία συναπόφασης. Καλό θα ήταν να έχουμε μια ευρωπαϊκή σύνολη προσέγγιση στο σύστημα αξιολόγησης του Σέγγεν και περιμένω έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον τη νέα σας πρόταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μποσκούρτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την εισαγωγή σας. Ε, πάρα πολλά θέματα καλύψατε, μικρά μεν, αλλά σε ορισμένα θα ήθελα λίγο να παραμείνω και να ζητήσω περισσότερη ενημέρωση. Χαίρομαι πολύ που είπατε ότι για την απελευθέρωση ε, των θεωρήσεων για τη Βοσνία και την Αλβανία επίκειται. Δεν έχω δει ακόμα ε, την πρόταση. Είπατε ότι θα στο φθινόπωρο αλλά η έκθεση των εμπειρογνωμόνων ε, έχει πάρει το πράσινο φως. Ε, θα μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο σε αυτό. Ε, κάτι άλλο. Είπατε για πολλές χώρες, Μορδαβία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν και πάει λέγοντας που σας απασχολούν. Με την Τουρκία τι γίνεται που είναι χώρα υποψήφια προς ένταξη. Ακούμε πολλά, ακούμε για συμφωνίες επανεισδοχής γίνονται ολόκληρα ταξίδια προς την Τουρκία. Πώς έχει η κατάσταση των πραγμάτων εκεί. Και μια τελευταία ερώτηση. Κάποια στιγμή είπατε ότι το σύστημα αυτό οικονομικού εντοπισμού των τρομοκρατών TFTP βοήθησε να πιαστούν τρομοκράτες. Με οδήγησε λέει σε μεγαλύτερη ασφάλεια. Μπορείτε να μας δώσετε κανένα παράδειγμα πώς αυτό έγινε μέσω των οικονομικών στοιχείων. Ο κύριος Γιακολίνο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, μεγάλη ευχαρίστηση που σας συναντάω. Πάντα σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή, διότι όλα όσα μας λέτε είναι πάρα πολύ επίκαιρα και εύστοχα. Μεταξύ των προτάσεων που αναφέρατε, είναι η οδηγία για την ανταλλαγή και μετάθεση εργαζομένων μεταξύ επιχειρήσεων και για τους εποχιακούς εργαζομένους και η κοινωνική προστασία των εποχιακών εργαζομένων από, τρίτε, εργαζομένων από τρίτες χώρες. Πρόκειται για μια απάντηση στις απαιτήσεις που έχουν προβληθεί μέχρι τώρα και σωστά τοποθετηθήκατε. Πριν από λίγο Μιλήσατε για τη δυνατότητα που υπάρχει για την υποβολή σχεδίων πιλότου για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και μέσα από σχέδια πιλότου. Εμείς συναντήσαμε τον διευθυντή σας στο Μαν Σερβίζη λίγο πριν φύγουμε για τις διακοπές και συζητήσαμε ένα θέμα, συμφωνία, ένα θέμα σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης για τον επαναπατρισμό και την λογική ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών συνδέοντας αυτές τις ροές και με τις ανάγκες εργασίας. Και ο διευθυντής σας μας είπε ότι θα πήγαινε στη Λιβύη εκείνη την περίοδο και θα είχε και άλλες συναντήσεις διότι η Λιβύη όπως είναι γνωστό έχει μία σύμβαση συνεργασίας, μία συμφωνία συγγνώμη, συνεργασίας με την ε, Ιταλία. 39 για να είμαστε και πιο ακριβείς συμφωνίες έχουμε με τη Λιβύη. αλλά εμείς ε, θεωρούμε ότι πέρα από αυτές τις 39 συμφωνίες που έχουμε εμείς θα ήταν καλό να έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα ορίζεται από την Κομισιόν για αυτά τα θέματα που θα ρυθμίζουν και ορισμένες ε, ε, εφαρμοστικές λεπτομέρειες βέβαια. Τώρα οι ροές ε, αλλάζουν. Παλιά ερχόντουσαν με σχεδίες ε, στη Λαμπεντούζα. Τώρα έρχονται με γιώτη με την λαθρομετανάστες. Έχουν αλλάξει λοιπόν τα επίπεδα των ροών και το στυλ αυτής της ροής. Ρωτώ λοιπόν, υπάρχει μια κάποια συγκεκριμένη δυνατότητα αυτές οι διμερείς ε, συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών Υπάρχει περίπτωση λοιπόν αυτές οι διμερείς συμφωνίες να υποκατασταθούν από συμφωνίες που θα προσυπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μούλτερ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Επίτροπο που ήρθε εδώ. Έχω την έντονη εντύπωση ότι είναι ειλικρινή όταν λέει ότι θέλει να έχει ανοιχτό διάλογο και διάβλο επικοινωνία με το Κοινοβούλιο. Ερωτήσεις δύο έχω. Η πρώτη έχει να κάνει με το πακέτο ασύλου. Από ό,τι κατάλαβα από προηγούμενη απάντηση που δώσατε θα έρθει πριν τις 20 Δεκεμβρίου, άρα έχω καλυφθεί. Δεύτερη ερώτηση, επειδή είμαι νέο μέλος εδώ σε αυτή την Επιτροπή, μπορεί να είναι ανόητη ερώτηση χρόνια ολόκληρα. Μιλάμε για ένα Ευρωπαίο εισαγγελέα. Ε, με τη συνθήκη της Λισαβόνας τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τι γίνεται, κινείται τίποτα προς την κατεύθυνση αυτή. για να ε, αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. ε, Ευχαριστώ κυρία Μαλστρόμ. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Λυπούμε που δεν άκουσα το πρώτο τμήμα της τοποθέτησής σας, αλλά θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω το εξής, να σας θέσω δηλαδή μια προτεραιότητα. Πιστεύετε ότι, αξίζει τον κόπο να μελετηθεί το θέμα της βίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η βία που υπόκεινται οι γυναίκες μόνο για το γεγονός ότι είναι γυναίκες. Πρόκειται για μια σιωπηλή βία, διότι ανήκει στην ιδιωτική ε, σφαίρα, στον ιδιωτικό βίο και χάνονται τα ποσοστά αυτής της βίας μέσα στα γενικά ποσοστά ε, ε, φόνων. Θα ήθελα λοιπόν εμείς να προσέξουμε αυτούς τους θανάτους που μπορούμε να αποφύγουμε γιατί ναι μεν μπορούμε να λέμε ότι πολλοί οφείλονται από αυτούς τους θανάτους ε, στη διαφορετική κουλτούρα ε, αυτό όμως ε, αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει στη δική μας κουλτούρα και θα έπρεπε να μπορέσουμε να μετρήσουμε αυτούς τους, αυτούς τους θανάτους. Η Ισπανία έχει δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο σχετικά θα ήθελα να ξέρω μέσα από τις ε, κοινέ δολοφονίες ποιες είναι οι χώρες εκείνες που ανασύρουν τα συγκεκριμένα στοιχεία για τις δολοφονίες γυναικών. Διότι έχουμε στοιχεία, ε, μας λείπουν στοιχεία. Εμείς όμως στην Ισπανία έχουμε 44 φόνους ένα χρόνο. Κάθε τρεις ε, μέρες στη Γαλλία δολοφονείται μία γυναίκα. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει όμω δεν έχουν ακριβή στοιχεία. Κατά την Ισπανική Προεδρία έγινε μία πρόταση σχετικά και βρισκόμαστε στη, ακόμη στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Αλλά συμβαίνει το εξής παράδοξο. Στα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις Υπάρχουν. Κοιτάξτε, έχουμε δύο διακόπτη την πρότασή της η ομιλήτρια και λέει εμείς έχουμε μία Ευρώπη δύο νο, ταχυτήτων μέσα στην ίδια ενόμη τάξη. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πρόληψη για αυτό του είδους ε, την εγκληματικότητα. Αυτό λέει η Κομισιόν. Εγώ όμως δεν το βλέπω διότι η πρόληψη εξαρτάται από τις διαφορετικές αρχές οι οποίες εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. Οι αρχές λοιπόν που ασχολούνται με τα εσωτερικά θέματα θα μπορούσαν να εργαστούν στην πρόληψη, δηλαδή ξεκινώντας εκείνη τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην αποφυγή του εγκλήματος. Η αστυνομία, οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα. Κοιτάστε, για την, παιδοπορνογραφία Υπάρχουν μέτρα για την πρόληψη, κλείνουμε τις σελίδες ίντερνετ, αλλά η αστυνομία ή ο δικαστής μπορούν να παρέμβουν. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κάτι το αντίστοιχο, διότι οι δολοφονίες γίνονται στο μεταξύ. Θα ήθελα να το διαβιβάσετε αυτό και στην Επίτροπο, την κυρία Ρέντινγκ, που ασχολείται με τη δικαιοσύνη, για να βρούμε μια λύση.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 See. Now the floor back to Commissioner Malmström. Επανερχόμαστε τώρα στην Επίτροπο, κυρία μας. Θα είμαι σύντομη, κύριε Πρόεδρε, απαντώντα όμω σε κάθε ερώτηση. Κυρία Ινθενβέλτ, όπω είπα και στην αρχή, το είχα διαβάσει το θέμα σήμερα το πρωί στη Μοντ και μου έδωσε και η κυρία Βεζιά σήμερα το πρωί κάποιο υλικό να διαβάσω. Βεβαίω είναι ανησυχητικό το θέμα και θα το συμπεριλάβουμε στην έρευνα που έχει ξεκινήσει η Κομισιόν υπό την ε, κυρία Ρέντινγκ, την Αντιπρόεδρε, αλλά βεβαίως ε, με την εμπλοκή και πολλών άλλων επιτρόπων, γιατί το θέμα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Και βεβαίως θα ε, μελετήσουμε και αυτό που λέει η κυρία Βερζιά. Ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα να απελάσει άτομα εάν διαπράξουν αδικήματα στο εδαφός του. Αλλά εδώ έχουμε το θέμα αν υπάρχει εξατομικευμένη διαδικασία, αν υπάρχει ενημέρωση, αν δεν πρόκειται για μια συλλογική κίνηση. Ε, αυτό θα μελετήσουμε και θα το ε, συζητήσουμε ως προς τη... Για το PNR, βεβαίως, ναι. Ευχαριστώ για την υπομονή ε, του Κοινοβουλίου επί του θέματος. Η Κομισιόν την Τρίτη στο Στρασβούργο θα εγκρίνει μια ανακοίνωση και όπως σας είπα θα συναντηθώ μαζί σας για να εξασφαλίσω ότι δεν θα υπάρξει κανένα λάθος και ότι δεν θα φύγει από την ημερήσια διάταξη κατά κάποιο τρόπο. Θα σας αναμερώσω άμεσα για αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει πριν ενημερώσω φυσικά και τον τύπο. Εσείς πρώτα. Όσον αφορά την ερώτησή σας για το ε, ευρωπαϊκό PNR, ε, είναι ενδιαφέρον το θέμα, ε, θα το μελετήσω. Για το ΣΥΣ, ναι, το βασικό θέμα κύριε Πολού είναι ότι έχω μια κοινή αξιολόγηση του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Το, η πρώτη ημερομηνία επετεύχθη σωστά. Ε, διαπραγματευόμαστε με τον ανάδοχο για τις λεπτομέρειες και το τίμημα και θα υπάρξει ε, έγγραφο ε, την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Θα υποβληθεί στο Συμβούλιο Τζάι, θα υπάρχει διαδικασία, ο προπολογισμό και φυσικά θα, εκ των υστέρων το έγγραφο αυτό θα έρθει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προετοιμάζουμε και τη δεύτερη σημαντική ημερομηνία όπου θα γίνει η τελική δοκιμασία και ελπίζουμε ότι θα είναι επιτυχής και θα τεθεί εν Αλλά τα τελικά στοιχεία θα υπάρχουν το ε, Οκτώβριο. Για το ΒΙΣ, όπως ξέρετε και εσείς, υπάρξει, έχει υπάρξει καθυστέρηση. Θα ζητήσω από τις υπηρεσίες μου να σας ε, στείλω μια πλήρη επιστολή για το πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε για να υπάρχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και εξ όσων γνωρίζω είμαστε, ε, προετοιμαζόμαστε για θέση ενισχύ τον Ιούνιο του 2011. Για το σύστημα αξιολόγησης του Σέγγιν έγινε επί του θέματος συζήτηση ε, στο Κοινοβούλιο, όχι πολύ παλιά, η Κομισιόν σαφώς πιστεύει ότι πρέπει να συμμετάσχει. Για την κυρία Περσκούτ. Ναι, υπάρχει έκθεση, ανάλυση εμπειρογνωμόνων, την οποία θα σας στείλουμε στο Κοινοβούλιο δηλαδή σήμερα, θα υπάρχει αξιολόγηση εκεί. Εκεί βλέπουμε ότι έχει σημειωθεί σοβαρή πρόοδος και στις δύο χώρες για όλα τα κριτήρια ε, που έχουν τεθεί και έχουμε ε, δώσει μια προσωρινή καταφατική απάντηση από την Άνοιξη ε, και βεβαίως συνεχίζει το πράσινο φως κομισιόν, το συζητάμε, ε, θα το συζητήσουμε με το Συμβούλιο μέσα στο φθινόπωρο και φυσικά με το Κοινοβούλιο και ξέρω ότι μπορώ να υπολογίσω την υποστήριξή σας. Επί της Τουρκίας τώρα δεν έχουμε ολοκληρώνεται μία ε, συμφωνία επανεισδοχής με την Τουρκία. Υπάρχουν λεπτομέρειες που πρέπει να δούμε. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να υπάρξει. Οι τουρκικές αρχές συνεργάστηκαν και ήταν πολύ επικοδομητικές. Δεν έχει συνδεθεί, όπως σε άλλες περιπτώσεις, συνδεθεί με την ελευθερία των θεωρήσεων διαβατηρίων ε, αλλά εκ των υστέρων, αφού ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, η Κομισιόν θα ήθελε να ξεκινήσει ένα διάλογο με τι τουρκικέ αρχέ επ' αυτού. Φέτο το καλοκαίρι έγινε μια συνάντηση σε επίσημο επίπεδο για το πώ μπορεί να εφαρμοστεί ο νέο κώδικα θεωρήσεων, πράγμα που θα, θα διευκολύνει του ε, πολίτε τη Τουρκία ε, στι διαδικασίε ε, του και ελπίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα διάλογο επ' αυτού, όχι, που μάλιστα να μην καθυστερήσει πολύ. Για το TFTP, όπως είπα και τους δύο προηγούμενους ερωτώντες, Παραδείγματο χάρη, η, ομάδα, η τρομοκρατική ομάδα που σταματήσαμε στην Νορβηγία, ε, σταμάτησε χάρη στο SWIFT, τα στοιχεία TFTP. Χρήσιμο. Κύριε Τζακολίνο, βεβαίως, θεωρώ ότι είναι πάντοτε καλύτερο να υπάρχει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τους γειτονές μας, Λιβύη και άλλες χώρες της Μεσογείου. Γίνονται αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με πολλές χώρες επί πολλά χρόνια. Η Λιβύη είναι χώρα δύσκολη όπως γνωρίζετε, αλλά σημαντικός γείτονας. Γι' αυτό προσεγγίσαμε τις λιβικές αρχές. Έχω ξεκινήσει διάλογο μαζί τους για να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε και να υπάρξει μια ε, ρύθμιση η Ευρωπαϊκή Συμφωνία έχει το πλεονέκτημα ότι είναι διαφανής για όλους. Μπορούμε να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα σχετικά, όχι μόνο μεταναστευτική πολιτική, αλλά και το εμπόριο, ε, συνεργασία, ανθρώπινα δικαιώματα. Προσεγγίζουμε λοιπόν τις λιβικές αρχές και αν το καταφέρουμε ε, σκοπεύω να τους επισκεφθώ φέτος το φθινόπωρο για να επιτευχθεί μαζί τους μια συναυθή, μια Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Κύριε Μουλίτερ, δεν υπάρχουν βλακώδεις ερωτήσεις, υπάρχουν βλακώδεις απαντήσεις μόνο στην πολιτική και ε, κατόπιν αυτού ελπίζω ότι η δική μου απάντηση δεν θα είναι ε, βλακώδης. Ε, ο Γενικός εισαγγελέα είναι αμφιλεγόμενο θέμα στα κρατημέλη, ακόμα και αν υπάρχει. Είναι θέμα ευθύνη της κυρίας Ρέντινγκ, η οποία συζητά στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης ε, ε, το θέμα. Είναι δύσκολο να επέλθει η συμφωνία. Προβλέπει όμω η Κομισιόν ε, την θέση της ενισχύ. Θα χρειαστεί όμω κάποιος χρόνος γιατί δεν υπάρχει ομοφωνία. Προς την κυρία Συμφωνώ. Συμμερίζομαι τη δική σας αφοσίωση να κάνουμε κάτι για αυτό το θέμα. Είναι τρομακτικά αυτά που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εμπόριο γυναικών, η διακίνηση λευκής αρκός είναι πάρα πολύ φρικτό και απαράδεκτο ε, θέμα, αλλά επίσης απαράδεκτο είναι και το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Και είναι λυπηρό να βλέπουμε πόσους αφορά αυτό και στη χώρα τη δική μου, φανταστείτε, είναι τόσο ε, σοβαρό αυτό το πρόβλημα. Ανταλλαγή απόψεων, ναι, βεβαίως πάντα ε, βοηθάει, αλλά σε τελική ανάλυση η ευθύνη είναι στα κράτη-μέλη. Θα διαβιβάσω την ισχυρή σας έκκληση προς τη συνάδελφό μου, την κυρία Ρέντινγκ, που προετοιμάζει ένα έγγραφο για την ισότητα των φύλων. Θα ε, σας πω τι κάνετε, τι ε, θα μου πει απαντώντας τα όσα είπατε. Αυτά νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι απάντησα σε όλα τα στοιχεία, όχι με την ακριβή σειρά, επικαλύψει είχαμε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πάντα η συζήτηση μαζί σας είναι ενδιαφέρουσα και οι υπηρεσίε μου και εγώ είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας για να ε, συνεργαστούμε και στο μέλλον και το φθινόπωρο. Το ίδιο ισχύει και για μας. The same goes here. Νομίζω και είμαι βέβαιος ότι εκφράζω το αίσθημα ε, όλης της Επιτροπής ευχαριστώντας σας και δηλώνοντας και εμείς προθυμία να συνεργαστούμε. Έχουμε ε, πολύ καλή συνεργασία. Ε, έχει καθιερωθεί αυτή η πρακτική, πάρα πολύ καλή. Προσβλέπω και στο μέλλον να συνεχίσουμε ε, με αυτόν τον τρόπο, με αυτούς τους ρυθμούς να ανταλλάσσουμε απόψεις και να μας ενημερώνετε. Σας ευχαριστώ πολύ και περνάμε στο επόμενο θέμα. porque tema europeo. Porque es un tema Yes. Yes, Χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Ευχαριστήσαμε την Επίτροπο. Χαίρετε. Ε, περνάμε στο σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη. Συμφωνία προστασία δεδομένων μεταξύ της Ένωσης και των ΗΠΑ για σκοπούς επιβολής του νόμου. Εδώ πρόκειται για μια διμερή συμφωνία και θα μας ενημερώσει ο συνάδελφός μας, κύριος Άρμπρεχτ, εδώ παρόν, εισηγητής. Θα μας παρουσιάσει τα δύο πρώτα έγγραφα εργασίας μέσα στα επόμενα λεπτά για τη μελλοντική συνεργασία για τη Συμφωνία Προστασίας Δεδομένων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και είπα ΕΕ, ε, στα διάφορα στάδια μιας ποινική δίωξης ε, και ε, στα πλαίσια της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε θέματα ποινικά. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Άρμπρεχτ και μετά θα κάνουμε και μια μικρή συζήτηση για τα υπόλοιπα μέλη που θέλουν το λόγο. Θα ακούσουμε και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής και την Προεδρία του Συμβουλίου που παρευρίσκεται για το θέμα αυτό. Παρακαλώ, κύριε Άλμπρεχτ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Στα αγγλικά ο κύριος Άλμπρεχτ για την ευκαιρία που μου δίνετε για πρώτη φορά να σας μιλήσω εδώ για αυτή την τόσο σημαντική συμφωνία. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, την κυρία Ρέντινγκ και τις υπηρεσίες της για τις διευκολύσεις που μου παρήχαν και εμένα και τους και τους εισηγητές καθ' όλη τη διάρκεια της ε, διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για την εντολή. Εδώ και χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχει ζητήσει να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία ε, με ένα συνολικό πλαίσιο, πραγματικά συνεκτική και ε, πλήρης ε, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όταν μεταφέρονται σε θέματα επιβολής του νόμου, δικαίου και συνεργασίας στο ποινικό δίκαιο. Η συμφωνία αυτή θεωρείται δεσμευτικό πλαίσιο για όλες τις μεταφορές δεδομένων και το SWIFT και το PNR. Μάθαμε πρόσφατα ότι γίνανε σχετικές συζητήσεις και σύμφωνα με τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτομάτως αλλάζει έτσι και ο τρόπος με τον οποίο είχαμε μέτρα και ελπίζω να είναι πολύ ε, ε, πλήρης συνεκτική, συνοπτική συμφωνία Για το TNTP και για το SWIFT επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχουμε γενικές αρχές που να ε, μοιραζόμαστε με τη ΣΥΠΑ για την προστασία ε, σε θέματα ασφαλείας και ποινικέ υποθέσεις. Οπότε, θα ήθελα να σας πω ότι σε συνεργασία με τη Γραμματεία έχουμε εκπονήσει δύο πρώτα έγγραφα εργασίας. Πρώτο, για να δούμε τι ισχύει για την προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενός και στι ΗΠΑ αφετέρου. Και ε, ως βουλευτές ε, θα έχουμε έτσι μια κοινή βάση. Θα γνωρίζουμε ποιες είναι οι διαφορές μας, τι ισχύει και ποιες είναι και οι δυσκολίε που θα πρέπει να ε, ξεπεράσουμε για να συναντηθούν οι απόψεις μας για την προστασία των δεδομένων. Θα ήθελα να σας πω από την αρχή ότι αυτά τα δύο είναι μόνο τα πρώτα έγγραφα, είναι έγγραφα εργασίας. Ε, έπονται άλλα δύο ε, τις επόμενες εβδομάδες για θέματα περιεχομένου και μορφής της συμφωνίας αυτής. Δεν είμαστε ακόμα ε, σε στάδιο που να μπορούμε να συζητήσουμε σε λεπτομέρειες στην ουσία. Ε, προς το παρόν μιλάμε ακόμα για την εντολή του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Γι' αυτό έχουμε λοιπόν τα έγγραφα αυτά εργασίες και έτσι τα χαρακτηρίζουμε για το γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ και έχουμε δύο βασικές διαφορές για τον κοινοτικό νόμο, η ιδιωτική σφαίρα και η προστασία των δεδομένων είναι ρητά αναγνωρισμένα θεμελιώδη δικαιώματα. Στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και στο άρθρο 8 συγκεκριμένα ε, και στο 7 και στη Νέα Συνθήκη, στο άρθρο 16, αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα και ρητά ορίζεται ότι αυτό το θέμα είναι ε, θεμελιώδες δικαίωμα. Ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες αυτό δεν θεωρείται κλασικό θεμελιώδης δικαίωμα, αλλά κάτι που μπορούν με αυτονομία να αποφασίζουν. Και ότι υπάρχει έτσι μια λελογισμένη ε, ελπίδα ή ε, προσδοκία για προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ας πούμε υπάρχει ο νόμος Privacy Act του 1974 ε, για την αρχή της δίκαιης και σωστής ενημέρωσης είναι θέματα και υποκειμενικά για το ποιος έχει πρόσβαση βέβαια. Αλλά στην Ευρώπη έχουμε ένα είδος ελαχιστοποίησης των ε, προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται. Αυτό δεν το θεωρούν σκόπιμο οι Αμερικανοί. Και επίσης περιορίζεται σαφώς ο στόχος και ο σκοπός. Αλλά και αυτό δεν αναφέρεται τόσο ρητά στην ε, Αμερικανική νομοθεσία. Και κάτι άλλο. Είναι γενική διαφορά. Είναι ανεξάρτητες αρχές ε, προστασίας ε, δεδομένων στην Ευρώπη, ενώ στις Ηνωμένε Πολιτείες πρόκειται για γραφεία για υπηρεσίες εντός των θεσμών. Δεν υπάρχει δηλαδή ε, επόπτης ε, προστασίας πολιτικών δεδομένων ανεξάρτητος. Αυτές είναι οι διαφορές μας και όπως γνωρίζουμε και από τη συμφωνία TFTP και PNA όταν πρόκειται για προσφυγή σε δικαιοσύνη ε, υπάρχουν διαφορές και προβλήματα, κυρίως για πολίτες που δεν είναι Αμερικανοί. Τα ξέρει αυτά η κυρία Ρέντιν και θα πρέπει να τα λάβει υπόψη της στις διαπραγματεύσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει μια νομοθεσία ο πρώην τρίτος πυλώνας για θέματα αστυνομική συνεργασίας και εσωτερικών. Αλλά δεν είναι μόνο το τρίτο πυλώνα, γιατί υπάρχουν ειδικέ ρυθμίσεις για την Ευρωπόλ, για τη σύμβαση του ΠΡΟΥΜ και κάτι διμερεί συμβάσεις και τώρα την TFTP και PNR με ειδικέ διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. θα πρέπει να είναι συνολική και αυτή η οδηγία για τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και επίσης θα πρέπει αυτή η συμφωνία πλαίσιο να αποτελέσει ένα γνώμονα, ε, ένα μπούσουλα που θα μας οδηγεί και σε επόμενες συμφωνίες. Πάντα ε, για θέματα τρίτου πυλώνα ε, θα πρέπει να είναι αντίστοιχη ας πούμε τη συμφωνία Safe Hub για τον ιδιωτικό τομέα. Κάτι άλλο που θα πρέπει να διευκρινιστεί τις ερχόμενες εβδομάδες και μήνες και νομίζω ότι αυτό θα το συμπεριλάβω στα επόμενα έγγραφα εργασίας είναι το πεδίο εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Δηλαδή, Πώς συνδυάζουμε αρχές όπως είναι η αναλογικότητα που αλλιώς αντιμετωπίζεται στην Ευρώπη και αλλιώς στο Αμερικανικό δίκαιο και πώς ξεπερνούμε τα προβλήματα διαφορετικών ε, ρυθμίσεων όταν ε, γίνεται λόγος για ελεγχιστοποίηση των στοιχείων ε, ή τι ισχύει για την αμοιβαιότητα και πώς αντιμετωπίζουμε τα θέματα διαφάνειας ή προστασίας των αρχών και των ανεξαρτήτων αρχών. Πέρα από το περιεχόμενο θα πρέπει να συζητήσουμε και τη μορφή της συμφωνίας, γιατί και αυτό απασχολεί τα έγγραφα εργασίας που δεν οριστικά όπως σας είπα. Η ευρωπαϊκή πλευρά της διαπραγμάτευσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτιμάει δεσμευτική ε, μορφή συνεργασίας, όπως είναι η Διεθνή Συνθήκη για παράδειγμα. Αυτό ε, σημαίνει ε, στις ΗΠΑ ενέχεται εκεί και το Κογκρέσο. Θα πρέπει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν, πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα. Εμείς θέλουμε να έχουμε δεσμευτικούς στόχους κατέρωθαν του Ατλαντικού. Και αυτό μπορεί να σημαίνει αλλαγή νομοθεσίας και στις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη. Αυτά για το περιεχόμενο του εγγράφου εργασίας ή των δύο εγγράφων συμφωνήσαμε τους κοιόδης ηγητές από κοινού να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και να γίνει και ακρόαση εδώ στην Επιτροπή μας. Θα βρούμε πότε με τη γραμματεία. Τέλειο Οκτωβρίου κάπου. Και επίσης να γίνει μια αντιπροσωπεία, έχει αποφασιστεί αυτό για τη συμφωνία αυτή, αλλά όχι πριν τα τέλη του έτους. Ε, μια αποστολή δηλαδή εκεί, κάπου στις αρχές του επόμενου έτους. για να συνεργαστούμε στενά με τους συναδέλφου μα στο Κογκρέσο και τη Γερουσία. Αυτό άλλωστε είχε αποφασιστεί και στι διαπραγματεύσεις για το TFTP. όπου ζητήσαμε από τον πρόεδρο Μπούζεκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουμε κάποιο είδου συνεργασία με τον Κογκρέσο για την προστασία των δεδομένων. Για να τελειώσω, Σα λέω είναι ανεξελίξια ε, η διαδικασία. Η εντολή δεν πρόκειται να εγκριθεί πιστεύω πριν από το τέλη Νοεμβρίου. Προλαβαίνουμε λοιπόν να βγάλουμε μέχρι και ψήφισμα ή σχέδιο ψηφίσματος της Επιτροπής μας για τη Σύνοδο Ολομελίας του Νοεμβρίου στο Στρασβούργο, έτσι ώστε εμείς και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Για την εντολή εγκαίρως. Παρακαλώ τα σχόλιά σας και θέλω πραγματικά να έχουμε άλλη ενημέρωση ε, και να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας και για τη συμφωνία και για τα έγγραφα εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Βεβαίω και θα γίνει συζήτηση. Βλέπω ήδη οι μέλη που έχουν ζητήσει το λόγο. Προηγουμένω όμω, καλύτερα θα ήταν να ακούσουμε την άποψη τη Κομισιόν και μετά του Συμβουλίου. Η κυρία Μπουλανζέκ, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Μπουλανζέκ. Monsieur le Président. όπως είπε και ο εισηγητής, η Κομισιόν στα τέλη Μαΐου του 2010 έκρινε μία σύσταση προς το Συμβούλιο που ε, επιτρέπει, επιτρέπει την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑ για το θέμα μεταφοράς ε, δεδομένων ε, για την αποφυγή ποινικών ε, θεμάτων. Και επίσης και δικαστικές πληροφορίες σχετικά με ποινικέ διαδικασίες. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει και συζητώνται στο Συμβούλιο. Να σας θυμίσω τους τέσσερις βασικούς στόχους ε, της Κομισιόν σχετικά με την παρουσίαση αυτής της σύστασης. Πρώτο, η συμφωνία θα πρέπει να εγκιάται στο μάξιμουμ την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών των ατόμων και κυρίως της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και αυτό σύμφωνα με την ε, Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη Συνθήκη της Λισαβόνας για την ανταλλαγή δηλαδή πάντα των δεδομένων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για την επιβολή του νόμου. Δεύτερο, νομικό πλαίσιο δεσμευτικό για την προστασία των δεδομένων στα πλαίσια των ανταλλαγών που ανέφερα. Στόχος είναι να αποφύγουμε αβεβαιότητες και κενά που αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν και αυτό λόγω ε, των διαφορετικών πρακτικών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα προστασίας δεδομένων. Τρίτο, η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων όταν αυτά τα δεδομένα μεταφέρονται και εξετάζονται στις ε, διάφορες χώρες. Θα πρέπει εμείς όταν εξετάζουμε αυτά τα ποινικά και δικαστικά θέματα θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μέσα στα πλαίσια της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, στα πλαίσια των ποινικών υποθέσεων. Θα πρέπει λοιπόν να έλεγα να λαμβάνουμε υπόψη την προστασία των προσωπικών στοιχείων. Και δεν θα υπάρχει εξαίρεση. Εμείς ε, δεν προτείνουμε να... Εμείς ε, δεν θέλουμε να αλλάξουμε ή να καταργήσουμε μία νομική βάση. Έχουμε βέβαια το προηγούμενο εμείς ε, της νομικής βάσης ε, για την ε, σχετική οδηγία 9546 όπου προβλέπεται μία νομική βάση αλλά δεν έχει να κάνει με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατικών φορέων. Ο κύριος Μωρό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Εγώ εδώ και 18 χρόνια ασχολούμαι με την προστασία των δεδομένων και ασχολήθηκα με το SWIFT και την μεταφορά ε, στοιχείων των επιβατών. Εργάζομαι ε, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ασχολούμαι με δικαιώματα του ανθρώπου. Πρόκειται για ένα ντοσιέ το οποίο γνωρίζω αρκετά καλά διότι μία από τις ε, δυσκολίες που έχουμε σε αυτού του είδους ε, τις υποθέσεις είναι να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το Αμερικανικό δίκαιο. Όπως πολύ σωστά το επισημαίνουν ε, οι νομικοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Αμερικανικό δίκαιο είναι ένα σύνθετο μοσαϊκό. Πρέπει λοιπόν καταρχήν το Συμβούλιο να συμφωνήσει για την εντολή και αυτό βάσει των στόχων που προτείνει η Κομισιόν και λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πρώτο βήμα της Ευρώπης προς τις Ηνωμένε Πολιτείες και των Ηνωμένων Πολιτείων προς την Ευρώπη ήταν οι στόχοι που, προσεγγίστηκαν από την συνεργασία της ε, Επιτροπής Στελεχών για την Προστασία Δεδομένων. Είναι σαφές ότι το, το αμερικανικό νομικό σύστημα και το δικό μας ε, δεν είναι ταυτόσημα. Αλλά μέσα στα πλαίσια της προστασίας δεδομένων στην, ε, στη High Level Data Protection Group Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας και στόχος μας σε αυτή τη φάση είναι να εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει το υπάρχον Αμερικανικό δίκαιο για να δούμε αν η προσφορά εγγύσεων επαρκεί και είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Εγώ θα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ε, να συνεργαστώ με τον κύριο Άλμπρεχτ και τους ε, σκιώδεις εισηγητές, διότι όλοι θέλουν, έχουμε τον ίδιο στόχο να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εφαρμογή αυτής της προστασίας στο Αμερικανικό Δίκαιο. Ευχαριστώ τα μέλη. Τώρα κάπου ε, ο κύριο Μπρόνς ότι ζήτησε το λόγο, άλλος, για αυτό το θέμα. Ο κύριος Μπρόνς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση μόνο, που δι... μπορεί να έχει απαντηθεί, αλλά έχω φτάσει σε μια ηλικία που καμιά φορά ξεχνάω. Ποιες εγγύησεις υπάρχουν να εμποδι... ώστε να εμποδιστούν οι Ηνωμένε Πολιτείε να μεταβιβάσει πληροφορίε που έχει λάβει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλε χώρε ή τα συμπεράσματα τα οποία... στα οποία καταλήγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε με βάση τα ευρωπαϊκά στοιχεία σε άλλε χώρε. Δηλαδή, ανησυχώ ότι μπορεί να μεταβιβάσει πληροφορίε ή συμπεράσματα με βάση αυτά τα δεδομένα, α πούμε, προ χώρε τη μια, μια ε, χώρα τη Μέση Ανατολή ή ένα άτομο ε, για μια τέτοια χώρα που μπορεί να μην υποστεί καλή μεταχείριση βάσει αυτών των στοιχείων ή ο κίνδυνος να στοχευθεί ένα τέτοιο άτομο για να συλληφθεί ή να δολοφονηθεί από άλλες χώρες της περιοχής. Υπάρχουν λοιπόν εγγυήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μεταβιβάσουν αυτές τις πληροφορίες σε τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Κυρία Σίπελ. Πιστεύω ότι η σύντομη συζήτηση έδειξε από τώρα πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση. Βεβαίως τα ε, δικαϊκά συστήματα είναι πολύ διαφορετικά, όχι μόνο μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο εσωτερικό της Ένωσης. Δεν είναι ενιαία τα συστήματα δικαίου των κρατών μελών. Γι' αυτό μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Τώρα, ποιο είναι το δύσκολο. Ε, πέρα των τυπικών και επισήμων τέτοιων συστημάτων, θα έχουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη για να υπάρχει η δεδομένη ε, συνεργασία. θέλει ε, εχέγγυα ο κύριος Μπρος, δεν υπάρχει 100% εγγύηση. Όταν συνάπτω μια συνθήκη, ε, μπαίνω στον κίνδυνο να μην τηρήσει το ένα συμβαλόμενο μέρος τα υποσχεθέντα. Αν δεν το κάνουμε όμως αυτό, ας ξεχάσουμε την πολιτική μας δράση εν γέννη. Μπορεί να είναι διαφορετικά τα συστήματα δικαίου και τα διάφορα ε, ήθη και έθιμα, αλλά θα πρέπει να ε, γίνονται πάντα σεβαστά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων και των άλλων πολιτών. Γι' αυτό με χαρά περιμένω το τρίτο έγγραφο εργασίας του κύριου Άλμπερτ Αφού ανέλησε την αρχική κατάσταση θα περιγράψει και τα υπόλοιπα και ελπίζω η συζήτηση να είναι πάρα πολύ ε, θερμή αλλά και πάρα πολύ αντικειμενική γιατί τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει μόνο η συναισθηματική φόρτιση αλλά και μια ασφάλεια για τα δεδομένα τους. Ευχαριστώ. Thank you. Any... Ευχαριστώ. Άλλο μέλος που θα ήθελε να κάνει ερώτηση. Όχι. Κύριε Άλμπρεχτ, έχετε και πάλι το λόγο για να σχολιάσετε κάτι. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να θεσπίσουμε τις προτεραιότητές μας, κυρίως όσον αφορά το θέμα των τρίτων χωρών, Φερπίν, και συγκεκριμένους περιορισμούς, όπως επίσης και τη δυνατότητα να υπάρξουν δεσμευτικές αρχές και από τις δύο πλευρές και από τις, ε, εκ μέρους και των δύο εταίρων για να περιοριστεί η χρήση των δεδομένων που μεταβιβάζονται. Και αυτό είναι σημαντικό επειδή μιλήσαμε για το TFTP, το PNR. Επιμένουμε λοιπόν να υπάρξουν όλα αυτά ε, και άρα θα Χαιρόμουν να με, ακούσω την άποψή σας για το έγγραφο εργασίας, να ακούσω ιδέες για τα επερχόμενα έγγραφα εργασίας και ιδέες επίσης για το πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, αλλά φυσικά και με βάση μια κοινή προσέγγιση, κοινέ αρχές για να εξασφαλίσουμε διεθνή συνεργασία. Γι' αυτό προτείνω να προσπαθήσουμε να επισημάνουμε ως Επιτροπή και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις αρχές επί των οποίων θέλουμε να επιμείνουμε για, αυτές τις, ε, για αυτή τη μεταφορά δεδομένων, να προσπαθήσουμε να είμαστε ενωμένοι ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, με βάση αυτές τις αρχές στις διαπραγματεύσεις μας. Ευχαριστώ. Okay. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε, ίσως θέλει η Κομισιόν να προσθέσει κάτι στο Συμβούλιο. Αν όχι, αν όχι, κλείνουμε το θέμα αυτό τη ημερήσιας διάταξης και περνάμε στο επόμενο που είναι το τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, το 6, που αφορά την ε, οδηγία για τα δικαιώματα των υπόπτων που έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, τους, ενημέρωση για τα δικαιώματά τους. Θα ακούσουμε την Κομισιόν σχετικά με την πρόταση οδηγίας. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί το δεύτερο βήμα του οδικού χάρτη επί των δικονομικών δικαιωμάτων που ενέκρινε πέρυσι το Συμβούλιο και που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Μόλις ε, με ενημέρωσε η γραμματεία, λέει ο πρόεδρος, ότι η Κομισιόν, που πρέπει να πάρει και το λόγο για να κάνει την παρουσίαση του θέματος, δεν εκπροσωπείται ακόμα εδώ, γιατί ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα διαλυματάκι, 10 λεπτά, 10 λεπτά και μετά θα έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Dear colleagues, no further delay. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας μην καθυστερούμε άλλο. If you do not mind, we'll resume our work. Λοιπόν, να επαναλάβουμε τις εργασίες μας αν δεν έχετε αντίρρηση. υποφεληθούμε να, του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας, οπότε περνάμε στο σημείο 6 που προβλέπει η ημερήσια διάταξη, δικαίωμα ενημέρωση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, το δικαίωμα των των υποπτών να ενημερώνονται για τα δικαίωματά τους. Είναι σημαντικό στοιχείο του προγράμματος Χόλμη, ένα πρώτο βήμα το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούνιο φέτος με δικαίωμα μετάφρασης και διερμηνίας στις ποινικέ διαδικασίες. Θα θυμόσαστε, η συγγήτρια ήταν η Βαρόνη Λούτφορτ. Τώρα ήρθαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, η οποία ζήτησε μια ευρύτερη διαδικασία εγγυήσεων στις ποινικέ διαδικασίες. Ε, για μακρόν το ζητάμε αυτό ως Επιτροπή. και πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Υπενθυμίζω ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ δεν έχει ακόμα ορίσει τους συντάκτες του θέματος, είναι θέμα που θα συζητηθεί με τους συντονιστές. Όμως θα ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλώς ορίσατε, κύριε Σόνκα. Σόμκα. Έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, κύριε. κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που σας, ε, έβαλα, σας έκανα με περιμένατε. Προσπάθησα να έρθω στην ώρα μου, ε, στην ώρα που έλεγε το σχέδιο μερίσιας διάταξης, αλλά Είχα μόλι, βγει από το κτίριο, μόλις μου τηλεφώνησαν ότι είχατε εξαντλήσει το προηγούμενο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε τώρα. Θέλω καταρχήν να σα ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω δηλαδή την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και εσάς προσωπικά κύριε Πρόεδρε για την θερμή υποστήριξη που προσφέρατε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ε, του τριμερούς διαλόγου για το μέτρο Α που αφορά την το δικαίωμα στην ενημέρωση και τη μετάφραση. Ένα μέτρο, ε, ε, η σχετική οδηγία για το οποίο θα εγκριθεί σύντομα από το Συμβούλιο, ελπίζουμε το επόμενο δεκαπενθήμερο, αποτελεί σαφή ένδειξη ότι τα θεσμικά όργανα εργάστηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε ο δικός χάρτης να υλοποιηθεί. Είμαστε ιδιαίτερε ευγνώμονε και φυσικά προσβλέπουμε να συνεχιστεί το ίδιο καλό πνεύμα στι διαπραγματεύσει τα υπόλοιπα μέτρα. Το επόμενο μέτρο θα είναι το Β. Μια πρόταση επί του δικαιώματος ενημέρωσης. Η πρόταση έχει ήδη εγκριθεί επίσημα από την Κομισιόν τον Ιούλιο και υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατόπιν. Οπότε προσβλέπουμε στην έναρξη των διαπραγματεύσεων ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα υπό την ε, ικανή καθοδήγηση της Βελγικής Προεδρίας. Η πρόταση θα απαντήσει συγκεκριμένα στην πρόσκληση που αναφέρει ο δικός χάρτης που εγκρίθηκε το περασμένο Δεκέμβριο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η πρόσκληση ανέφερε ότι το μέτρο Β είναι το δεύτερο βήμα της όλης διαδικασίας. Θα επιδιώξουμε να εναρμονίσουμε δύο πλευρές αυτού του δικαιώματος στην ενημέρωση με το μέτρο αυτό. Το δικαίωμα του υπόπτου, δηλαδή αφορά δικονομικά δικαιώματα και αφετέρου αφορά τις κατηγορίες γιατί κατηγορείται δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και τα δύο δικαιώματα αναφέρονται ρητά, ε, περιλαμβάνονται ρητά ή έμεσα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων άρθρο 6 και στην ομολογία του ε, Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Όμως, Πολλές είναι οι διαφορές στην πρακτική των κρατών μελών, πώς εφαρμόζονται δηλαδή αυτά τα δικαιώματα στα κράτη-μέλη. Ε, έχει διαφορά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και αυτό ισχύει και για το είδος των πληροφοριών που παρέχεται στον άνθρωπο, για το χρόνο τον οποίο ε, παρέχεται και τις μεθόδους με τις οποίες παρέχεται η ενημέρωση αυτή. Η Κομισιόν θα προτείνει οι ύποπτοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, να ε, έχουν ένα δικαίωμα των ε, δικαιωμάτων τους, ένα κείμενο των δικαιωμάτων τους γραπτό. Το οποίο θα, ένα κείμενο το οποίο θα συνταχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πληροφορίες για τα δικαιώματα των υπόπτων που θα υποβάλλονται γραπτά. Θα προτείνουμε ένα πρότυπο Έχουμε προτείνει ένα πρότυπο ως παράρτημα της πρότασης, αλλά υπογραμμίζω ότι είναι ένα ενδεικτικό πρότυπο, ένα ε, μοντέλο που δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Θέλουμε όμως να βοηθήσουμε στην εφαρμογή αυτής της υποχρέωσης για να υπάρξει ένα γραπτό κείμενο που θα ε, προειδοποιεί τους υπόπτους γνωρίζοντας ότι μόνο περίπου τα μισά κράτη-μέλη έχουν, το έχουν εφαρμόσει στην πράξη. Περίπου 15 κράτη-μέλη δεν έχουν γραπτό τέτοιο, κανένα γραπτό τέτοιο κείμενο. Φυσικά τα κράτη-μέλη ε, μπορούν να το συμπληρώσουν το κείμενο αυτό με άλλα δικαιώματα τα δικαιώματα αυτή τη στιγμή είναι τέσσερα. Και επίσης υπάρχει δυνατότητα να μην χρησιμοποιηθεί αυτό το πρότυπο, αυτό το μοντέλο, αλλά το μοντέλο που ήδη υπάρχει. Επίσης ε, υπάρχει και σε πολλές γλώσσες, σε πολλά κράτη-μέλη το κείμενο υπάρχει σε 40-50 γλώσσες, σε άλλα με λίγες. Η ιδέα είναι ότι ο κάθε υποπτός που θα έχει, θα παραλαμβάνει αυτό το κείμενο με τη σύλληψή του στο αστυνομικό τμήμα, θα, μεταφρά, θα έχει από μας, μάλλον εμείς θα μεταφράσουμε το κείμενο αυτό σε 23 γλώσσες και οι γλώσσες αυτές ε, μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν. Τώρα, οι πληροφορίες για την υπόθεση περιλαμβάνονται στο κείμενο αυτό, δηλαδή θα υπάρχουν πληροφορίες για την κατηγορία, για το τι κατηγορείται σε κάποια κρατημέλη που, πράγμα που περιλαμβάνει επίσης και το δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελο της υπόθεσης, δηλαδή τις πληροφορίες ε, που έχουν οι αρχές ε, κατά του υπόπτου. Το δικαίωμα της ενημέρωσης για την κατηγορία θα συμπεριλαμβάνει και πρόσβαση το φάκελο, το δικαίωμα, το δικαίωμα δηλαδή να αποκαλυφθούν, να γνωρίζει ο υποπτός ε, τις πληροφορίες που έχουν εναντίον του οι αρχές. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι και, πάλι ότι αυτό το μέτρο εντάσσεται στην προσπάθεια της Επιτροπής να επιτευχθεί ένα ελάχιστο επίπεδο δικαιωμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν εφαρμόσει ένα ελάχιστο επίπεδο. Και θέλουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη να ενισχύεται και βεβαίως να εφαρμόζονται τα αμοιβαία μέσα αναγνώρισης. Ελπίζουμε ότι δημιουργώντας αυτά τα δικαιώματα ως ένα ελάχιστο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσουμε ώστε η δικαστική συνεργασία ε, θα λειτουργήσει καλύτερα με τον απαιτούμενο βαθμό εμπιστοσύνης και άνεσης δεδομένου ότι και οι εισαγγελείς και οι δικαστές και οι πολίτες πρέπει να απολαμβάνουν αυτή τη κατάσταση σε περίπτωση δίκης. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Κατά τα άλλα έχω ολοκληρώσει. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. κύριε Ξόγκα. Open now for... Και τώρα αρχίζει η συζήτηση. Διαρωτώ με το Συμβούλιο, η Προεδρία. Μήπως θέλετε να πάρετε τον λόγο. Ο κύριος... Θέλετε τον λόγο, κύριε... Oui, ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, η Προεδρία ευχαριστεί το Συμβούλιο για την ε, ευχαριστεί την Κομισιόν για την πρωτοβουλία της. Η πρωτοβουλία της Κομισιόν ήταν μια πρωτοβουλία την οποία προσδοκούσε ιδιαίτερα το Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε το ρυθμό και να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έγγραφο και να περάσει σύντομα τον Οκτώβριο στο Συμβούλιο Πρόκειται για ένα επικουρικό δικαίωμα διαδικοστικού χαρακτήρα. Για το Συμβούλιο βέβαια είναι πρόωρο να πούμε τι θα αποφασίσουμε, αλλά σε επίπεδο αρχών αποτελεί ένα κοινό κατόφλι για το δικαίωμα πληροφόρησης και Σε αυτήν τη φάση η πρόταση της Κομισιόν λειτουργεί καταλητικά. Θα ξεκινήσει η ομάδα εργασίας την επόμενη εβδομάδα και το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό θα προσπαθήσει να αποφασίσει για αυτό το μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας και θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό και ο διάλογος με το Κοινοβούλιο. Θα δούμε λοιπόν πότε θα μπορέσουμε να έρθουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι μέχρι τα τέλη της ε, χρονιάς θα καταφέρουμε να έρθουμε. Ευχαριστώ. Τα μέλη τώρα της Επιτροπής, η κυρία Σίπελ πρώτη. Ζητήσατε το λόγο. Όχι. Α, καλά. Ο κύριος Άρβεκ τότε. Um, Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλώς είναι σας. Ε, ο χάρτης και τα ελάχιστα ε, πρότυπα και προδιαγραφές που θέλετε για τις ποινικέ διαδικασίες. Ε, για το δικαίωμα τώρα του κατηγορουμένου να έχει ή του υπόπτου ενημέρωση και γραπτή. Να του κοινοποιούνται δηλαδή γραπτό τα δικαιώματά του. Έχω την εξής ερώτηση το δικαίωμα να παραμείνει κανείς σιωπηλός, να μην πει τίποτα δηλαδή. Θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την επιστολή και με ποιο τρόπο θα κοινοποιείται, αν υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή, να, ένας υποπτός να μην μπορεί να πει κάτι που θα χρησιμοποιηθεί εναντίον του, που να τον κατηγορεί. γιατί είναι και ένα δικαίωμα που καλύπτει η Ευρωπαϊκή ε, Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και μετά η πρόσβαση στην ενημέρωση. Είναι πολύ κρίσιμο και αυτό. Δηλαδή, βεβαίως να υπάρχει δεδομένη κάποια πρόσβαση, αλλά και η υπεράσπιση, ο συνήγορος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ε, πρόσβασης να τα λαμβάνει τα έγγραφα, όχι να το στέλνουν σε ένα ε, κρυφό δωμάτιο, να τα συμβουλεύεται και να ξαναφεύγει. Δεν ξέρω αυτό πώς θα γίνει. Εκφράζονται κάποιες απόψεις, αλλά έχουν αποκρισταλωθεί. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της. Θα ήθελα να πω καταρχά ότι φαίνεται να είναι πολύ σαφέστερη η διαδικασία αυτή από εκείνη που ακολουθήσαμε ε, στο πρώτο ντοσχέ για τα δικονομικά δικαιώματα, όπου δεν ξέραμε ακριβώς τι ίσχυε και ποιες προτάσεις έπρεπε να ακολουθήσουμε. Ε, ευχαριστώ που επιστρέψαμε στον κόσμο της ε, ομαλότητας, όπου κάνει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο την εξετάζουν. Είμαι βέβαιος ότι θα αξιολογήσει θετικά αυτή την πρόταση το Κοινοβούλιο, όπως άλλωστε έκανε και με τις προηγούμενες. Έχω και εγώ δύο ερωτήσει για την περαιτέρω ενημέρωση, που μάλλον χρειάζονται περαιτέρω ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν μου επιτρέπετε. Πρώτον, γίνεται λόγος για μια γραπτή επιστολή δικαιωμάτων. Αλλά είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλι ότι δεν θα είναι εναρμονισμένο το γράμμα δικαιωμάτων. Τι εννοεί ακριβώς μπορεί να μας το εξηγήσει, γιατί ποια είναι τα εμπόδια που βλέπετε να σας εμποδίζουν ακριβώς, να σας αποτρέπουν να έχετε τα ίδια δικαιώματα και την ίδια επιστολή που να κοινοποιείτε σε όλους τους υπόπτους που συλλαμβάνονται στην Ευρώπη. Σε όλες τις χώρες της Ένωσης δηλαδή. Ποιο είναι το πρόβλημα, οι ελάχιστες προδιαγραφές, για να μπορούν τα κράτη-μέλη να προσθέτουν και άλλα δικαιώματα. Ή μήπως ακόμα και η ε, δυνατότητα επιβολής ε, γραπτών δικαιωμάτων του υπόπτου. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό. Δεύτερον, ποια θα είναι αυτά τα δικαιώματα. Μπορείτε να μας ε, δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Επιπλέον των όσων ρώτησε ο συνάδελφος Άλμπραχτ μόλις. Και γιατί να υπάρχει γραπτό κείμενο αντί για ανάγνωση ή εξήγηση. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και αγράμματοι ε, άνθρωποι, αναλφάβητοι ή μπορούν να ξέρουν να διαβάζουν αλλά δεν κατανοούν την επιστολή αυτή που τους διαβιβάζετε και τους υποβάλλετε με τα δικαιώματά τους. Αυτά. Ευχαριστώ. Thank you. Mrs. Ευχαριστώ κυρία Λούτφορντ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι η Ευρωβουλευτής που είναι υπεύθυνη για την ανώμαλη αυτή διαδικασία όπως ε, την περιέγραψε ο κύριος Σάιμον στη, προς το πρώτο φάση της ε, ε, δικονομικής, ε, των δικονομικών δικαιωμάτων. Χαίρομαι που ήρθε η απάντηση τόσο γρήγορα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά την, το μέτρο διερμηνίας και μετάφρασης, όπου είχαμε σοβαρές δυσκολίες σε σχέση με την θέση ενισχύτηση της συνθήκης Λισαβόνα. Ήμασταν κάπου στη μέση και δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Το καταφέραμε τελικά και χαίρομαι πολύ που αμέσως προχωρούμε. Ελπίζω ότι έτσι θα διατηρηθεί η όλη ε, ορμή και θα ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα δικονομικά μέτρα και αυτό είναι ένα ευχάριστο ξύπνημα μετά από μια περίοδο πενταετία στην οποία δεν κάναμε τίποτα για τα δικαιώματα αυτά. Είμαι πολύ ευγνώμων στην ομάδα των υπηρεσιών της Κομισιόν και στην ε, Αντιπρόεδρο κυρία Ρέντινγκ για την ε, όλη προσπάθεια αλλά και για, για το καλό αποτέλεσμα. Έχω λοιπόν μια ερώτηση και ελπίζω ότι στη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε αρκετά ε, σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία τουλάχιστον. Έχω μπερδευτεί λιγάκι, ίσως γιατί δεν έχω μελετήσει καλά τις εξηγήσει. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο άρθρο 3 και το άρθρο 4. Το άρθρο 3 αναφέρει τα δικαιώματα στην ενημέρωση όταν πρόκειται για κατηγορούμενο ή ύποπτο που πρέπει να ενημερωθεί προφανώς με μια απλή και αντιληπτή γλώσσα, ενώ όταν έχει συλληφθεί πρέπει άμεσα να ε, λάβει τα διαδικονομικά του δικαιώματα γραπτά. Είναι όμως απολύτως απαραίτητο να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στις δύο αυτές καταστάσεις. Δηλαδή, γιατί και ο ύποπτος να μην ε, παραλαμβάνει ένα πλήρες ε, κείμενο με τα δικαιώματά του. Γιατί υπάρχει αυτή η διακριτική μεταχείριση και οι πιθανές ε, περιπλοκές λόγω του ότι υπάρχουν δύο δυνατότητες. Θα ήταν πιο συνεπές, πιο συνεκτική η προσέγγιση και πιο ολοκληρωμένη η ενημέρωση αν το άρθρο 3 το απορροφούσε το άρθρο 4 και ότι αν τελικά καταλήγαμε σε μία και μόνη διαδικασία. Μία επιστολή, μία επιστολή με τα δικαιώματα. Thank you. Mr. Ευχαριστώ, Μπρόνς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξεπλάγιν που χρειάστηκε να πούμε στα κράτη-μέλη ότι τα οι ύποπτοι πρέπει να ενημερώνονται για το είδος των ουσιαστικών κατηγοριών αντίον και κυρίως για τα ελάχιστα δικονομικά δικαιώματα θεωρούσα ότι οι χώρες από μόνες τους θα είχαν τηρήσει αυτά τα ελάχιστα δικαιώματα. Αυτό που με ταράζει είναι ότι μπορεί οι άνθρωποι να μεταφερθούν σε αυτές τις χώρες με βάση ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης. Είχαμε επανειλημμένως πει ότι τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης θα μεταφέρουν ανθρώπους σε χώρες που δεν έχουν χειρότερα αποτελέσματα, αλλά τώρα βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται. Τουλάχιστον η συμφωνία για τα ελάχιστα ε, πρότυπα θα έπρεπε να είχε προηγηθεί ε, του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και όχι να, να έρθει χρόνια μετά. Ευχαριστώ κύριος Βαντεστόπ. Θα μιλήσω Ολλανδικά, λέει ο κύριος Βαντεστόπ. Στην πρόταση που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σελίδα 2 στα Ολλανδικά λέει ότι η οδηγία στις 8 ε, ε, Οκτωβρίου 2010 εγκρίθηκε για την διαρμηνία και τη μετάφραση για τους κατηγορουμένους. Περίεργο αυτό. Έχει διεγκριθεί στις 8 Οκτωβρίου. Επίσης αυτά που μας είπε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τα βρήκα πολύ συχνά. Ε, αυτά είναι θέματα επικουρικότητας. Μπορεί να μου το σχολιάσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν βρήκα πάρα πολύ στεναρή. Και το ποινικό δίκαιο παραμένει εθνικό, έτσι δεν είναι. Και βέβαια μπορούμε Ε, να έχουμε τη διεθνή εμπειρία και να ξέρουμε τι λέει ας πούμε το άρθρο 6 ότι έχει το δικαίωμα ο ύποπτο να τηρήσει τη σιωπή αλλά αυτά είναι θέματα που αφορούν τα κράτη, τα εθνικά κοινοβούλια και τη Βουλή της Ολλανδίας εδώ εσείς πώς θα τα συμπεριλάβετε θα τα ενημερώνετε, θα τα συμβουλεύεστε Μα είναι επικουρικότητα ε, αυτά τα θέματα και πώς θα εγγυηθείτε ότι δεν θα παραβιάσετε. Και το άρθρο 82 έχει να κάνει με διαφορετικές παραδόσεις και διαφορετικούς νομικούς πολιτισμούς στα κράτη-μέλη. Και επαναλαμβάνω ότι είναι θέμα επικορικότητας. Γιατί δεν μας τα λέτε αυτά. Και στην πράξη πώς θα το εφαρμόσετε. Ας πούμε, συλλαμβάνεται κάποιος. Θα του δώσω ένα φυλάδιο που υπάρχει σε 40 γλώσσες στο δικαίωμά του ή τι μπορεί να κάνει. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε πρακτικά πώς το φαντάζεστε αυτό. Ευχαριστώ. Okay. Καλώς, Πρόεδρος. Δεν θέλει άλλο το λόγο, δεν βλέπω άλλα χέρια. Α, είδα, η κυρία Ρωμέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα σηκώσει το χέρι μου, αλλά πιθανώς να μην με είδατε. Ίσως επειδή αυτή είναι και η πρώτη μου κοινοβουλευτική θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο, ήθελα να πω ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα φυσικά προβλέπουν ότι το δικαίωμα μετάφρασης και διερμηνίας είναι ένα πρωταρχικό δικαίωμα που σίγουρα θα πρέπει να προηγείται της δικές δίκης. Εμείς έχουμε το φιλοπορίας και το θέμα των δικαιωμάτων στο δικαστήριο θα πρέπει να συνεχιστεί. Είναι ένα πακέτο όλα αυτά. Δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε για δικαίωμα στη μετάφραση χωρίς το το... τη χάρτα των δικαιωμάτων και δεν μπορούμε να μιλάμε εμείς για χάρτα δικαιωμάτων αν δεν έχουμε όλα τα υπόλοιπα. Θα παρακαλούσα λοιπόν την Κομισιόν να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο στο θέμα των δικαιωμάτων και παρακαλώ και τη Βελγική Προεδρία να ενδιαφερθεί σχετικά διότι αν η Κομισιόν δεν λάβει την πρωτοβουλία τα κράτη-μέλη σε φάση κατεπήγοντος μπορούν αυτά να αναλάβουν το δικαίωμα πρωτοβουλίας. για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε εμείς αυτή τη χάρτα των δικαιωμάτων που να αποτελούν ένα μίνιμουμ για τους κρατούμενους στην Ευρώπη. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν η Κομισιόν έχει τη σχετική χαρτογράφηση με τα δικαιώματα των υπόπτων στις διάφορες χώρες Επίσης ε, θα θέλαμε να ξέρουμε πώς μπορούμε να μεσολαβήσουμε εμεί την επεξεργασία της ε, χάρτας και να ζητήσουμε από την Κομισιόν να μας ετοιμάσει κάτι το οποίο να είναι τουλάχιστον στο ελάχιστα αποδεκτό. Καλώς. Δεν έχουμε άλλους βουλευτές που να θέλουν το λόγο. Οπότε μπορούμε να επανέλθουμε στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Σόνκα, για ένα πρώτο γύρο σχολείων και απαντήσεων στις ερωτήσεις που σας έγιναν. Ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη για τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Αυτό είναι καλός ιονός για το πόσο ενδιαφέρον βρίσκεται το θέμα. Χαίρομαι και προσβλέπω στην ενεργό συμμετοχή σας στη διαδικασία συναπόφασης. Γιατί μόνο τα τέσσερα δικαιώματα στην επιστολή και όχι παραπάνω, ρωτήσατε. Επειδή σκοπός της Επιτροπής δεν ήταν να εναρμονίσει την ουσία του, του, της επιστολής δικαιωμάτων. Θέλαμε να δείξουμε προκαταρτικά ποια δικαιώματα πρέπει να υπάρχουν στην επιστολή δικαιωμάτων, αλλά στο επεξηγηματικό κείμενο ε, λέγεται σαφώς ότι είναι ενδεικτικό το κείμενο αυτό. Είναι μια ενδεικτική επιστολή, είναι ένα πρότυπο, μπορούν να το αλλάξουν, να το συμπληρώσουν και αυτό δεν θα επηρεάσει ε, ουδόλως τα υφιστά, τις, τις υφιστάμενες επιστολές δικαιωμάτων που χρησιμοποιούν τα κρατημέλη. Και δεύτερον, θέλουμε να ενημερώσουμε, να την επιστολή αυτή σε μερικά χρόνια όταν θα υπάρξει και η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας και τότε να προτείνουμε περαιτέρω δικαιώματα. Είναι απολύτως λογικό όταν έχουν εφαρμοστεί αυτά τα πέντε δικαιώματα του οδικού χάρτη που εγκρίθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη, τότε και τα πέντε δικαιώματα να περιλαμβάνονται στην επιστολή δικαιωμάτων. Μέχρι τότε το 2013-2014 πια μιλάμε. Μέχρι τότε έχει ολοκληρωθεί, που θα έχει ολοκληρωθεί ο δικός αυτός χάρτης θα μπορέπει να επανεξεταστεί το, η επιστολή δικαιωμάτων και τότε ίσως να γίνει υποχρεωτική γιατί μέχρι τότε θα, έχουν εναρμονιστεί, θα έχει εναρμονιστεί η ουσία αυτών των πέντε δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν να επιστρέψουμε σε αυτή την επιστολή σε μερικά χρόνια ε, τα 12 κράτη-μέλη που ήδη έχουν τέτοιες επιστολές δικαιωμάτων και τα χρησιμοποιούν στην πράξη, αναφέρονται ένα προς ένα στη μελέτη επιπτώσεων. Δυστυχώς δεν την έχω μαζί μου, θα μπορούσα να τα διαβάσω. Είναι όμως ένα δημόσιο έγγραφο, μπορείτε να διαβάσετε αυτή την επίπτωση, την αξιολόγηση των επιπτώσεων και θα δείτε ποια είναι τα 15 που δεν έχουν τέτοιου είδου επιστολή. Τώρα, αν είναι κάποιος αγράμματος ή έχει κάποιες ε, δυσκολίες. Η προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να υπάρχει βοήθεια για κάποιον που δεν μπορεί να καταλάβει ή να διαβάσει την επιστολή δικαιωμάτων. Άρα η επιστολή αυτή καθεαυτή πρέπει να είναι εύληπτη. Αν διαβάσατε το κείμενο που προσαρτάται στην πρόταση, δεν είναι πολύ ε, εξελιγμένο κανένα περίπλοκο νομικό κείμενο, είναι ένα απλό ξεκάθαρο κείμενο. Αν κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει τι λέει αυτό, μπορεί να δώσουμε και παραπάνω βοήθεια. Τώρα, οι διαφορές μεταξύ άρθρων 3 και 4. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορετική μεταχείριση ε, σε περίπτωση που μιλάμε για ύποπτο και σε περίπτωση που μιλάμε για άτομο που συλλαμβάνεται. Η διαφορά υπάρχει, προέρχεται από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, κατά των βασανιστήριων, τη CPT. Και υπάρχει στην έκθεση του 2009 αναφέρεται τα, ουσιαστικά... Ε, τα ε, πρότυπα της CPT, ένα ουσιαστικό κομμάτι της έκθεσης της CPT, όπου εξηγεί ότι οι υποπτοί που κυρίως χρειάζονται γραπτές πληροφορίες είναι αυτοί που συλλαμβάνονται, γιατί είναι πιο ευάλωτοι από αυτούς οι οποίοι ε, πρέπει να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ε, όντας ελεύθεροι, ε, χωρίς δηλαδή να έχουν τεθεί περιορισμό Και πάλι ίσως τελικά στο τέλος της διαδικασίας να συνδυαστούν οι δύο αυτές διατάξεις και να καταλήξουμε σε μια επιστολή δικαιωμάτων που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους. Ίσως τελικά στη συναπόφαση να έχουμε μια ε, επιστολή δικαιωμάτων που να χρησιμοποιείται για όλους τους υπόπτους. Μέχρι στιγμής ακολουθήσαμε, τηρήσαμε τον οδικό χάρτη και τη σειρά που προβλέπει αυτός. Και σκοπός μας είναι αυτή τη σειρά να την ακολουθήσουμε και στο μέλλον, γιατί θεωρούμε ότι η νομοθεσία τύπου Big Bang θα ξανααποτύχει. Το έχουμε ζήσει αυτό στο παρελθόν. Έχουμε προτείνει ήδη το 2004 ε, μια νομοθεσία τύπου Big Bang που πολλοί από εσά είχατε ζητήσει και η οποία πέτυχε διαφορετική συνθήκη τότε, διαφορετικές περιστάσεις ενδεχομένως, στο τρίτο τότε πυλώνα, αλλά και πάλι το γεγονός ότι χρειάστηκαν διαπραγματεύσεις για κάθε ένα από τα ε, διάφορα δικαιώματα οδήγησε την κατάσταση αποτυχία για διάφορους λόγους. Και θεωρήθηκε ότι ε, η αντιμετώπιση των δικαιωμάτων ένα προς ένα θα είναι το κλειδί για την επιτυχία. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ε, βαθμιαία προσέγγιση η οποία πιστεύουμε ότι θα μας οδηγήσει σε πλήρη εφαρμογή του δικού χάρτη. το τελευταίο ερώτημα. Ομολογούμε δηλαδή ότι θα έπρεπε τα δικαιώματα αυτά να έχουν εισαχθεί εδώ και πολύ καιρό όταν διαπραγματευόμασταν το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ε, και άλλα όργανα. Σαφώς αυτό είναι ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία των συμπερασμάτων του Τάμπερε πριν από 11 χρόνια. Οι αρχηγοί κρατών συνειδητοποίησαν ότι η αμοιβαία αναγνώριση δεν θα είχε αποτέλεσμα χωρίς να ε, υπάρξει προσπάθεια προσέγγισης των ελάχιστων προτύπων ε, μεταχείρισης των ανθρώπων και γι' αυτό συντάχθηκε μια πράσινη βίπλος, μια ουσιαστική πρόταση του 2004 η οποία πέτυχε και τώρα διαπραγματευόμαστε και πάλι με βάση τον οδικό χάρτη με την πλήρη δέσμευση των κρατών μελών της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα έχουμε μια, είμαστε σε μια εφεδρική λύση, δεν υπάρχει όμως άλλη και χαιρόμαστε που έχει ήδη εγκριθεί το μέτρο Α. Επανέρχομαι ε, στην ερώτηση του κυρίου Μπεζούτη που ε, διερωτήθηκε για την ημερομηνία στη σελίδα 2. Είναι η ημερομηνία ε, θέσπισης ε, έγκρισης που προβλέπεται για το μέτρο Α. Θεωρητικά είναι σωστή, έχει με 8 ε, Οκτωβρίου θα ε, εγκριθεί επίσημα το μέτρο Α. Δεν είναι η πρόταση, είναι το πρώτο ε, μέτρο στο οποίο αναφερόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Okay. Thank you. And maybe... Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο τίποτα, μήπως θα ήθελε να κάνει επιπλέον σχόλιο. Όχι, δεν χρειάζεται. Καλώς. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη για τη συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής μας. Παρακαλώ τους συντονιστές να παραμείνουν για να... Έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Μια που τελειώσαμε νωρίτερα όμω, θα πρότεινα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ενός τετάρτου για να έρθουν οι συντονιστές μας στις 6 ακριβώς, όπως είχε προβλεφθεί. Ευχαριστώ.